Okay. Ωραία. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Παρακαλώ καθίστε. Thank Σας κατευχαριστώ. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω καμία αντιρρήση. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι εγκρίνεται έγκριση των πρακτικών της 9ης Ιανουαρίου. Two meetings, 13th of January, 16th of January, 22nd to 23rd of January. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά, ως συνήθως αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Will be done tomorrow before votes. Uh, η ψηφοφορία οίκων Λίμπε αύριο το πρωί. Σας υπενθυμίζω ότι για τη μεταφορά των ποσών θα γίνει στις 9 στον αίθουσα της Λίμπε. 3 σε 50 και πρέπει μετά να επιστρέψουν τα μέλη σε αυτήν την αίθουσα, την 5G3, όπου θα αρχίσει η ψηφοφορία της οίκων στις 10. Πρώτα στη Λίμπε, μετά εδώ στην Ίκον. Γιατί από κοινού τα κάνουμε. Και το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, α, Πέμπτη, αύριο δηλαδή, και αυτό είχαμε πει να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη στις 22 Φεβρουαρίου στις 12.30. Αλλά από ό,τι κατάλαβα αυτό δεν βόλευε ορισμένους Δυστυχώς όμως δεν βρήκαμε άλλο τρόπο το Φεβρουάριο, μέσα στο Φεβρουάριο. Λοιπόν, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέβλημα βρωμίκου χρήματος όχι αύριο, αλλά την επόμενη Πέμπτη στις 12.30. Ίσως να σας φαίνεται περίεργος ο χρόνος, αλλά καλύτερα αυτό παρά το απόγευμα. Τώρα, το σημείο 4 και 5, γιατί προτείνω να τα δούμε κοινά διότι συνδέονται τα δύο θέματα. Αντί να πούμε τα πράγματα δύο φορές λοιπόν, να τα πούμε μία. Ο κάθε εισηγητής και σκιώδης θα λάβει το λόγο και φαντάζομαι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν πρώτα, ποιος είναι πρώτος είναι οι υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ο Γιώργος. Να υπενθυμίσω πως έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα οι δραστηριότητές μας και οι επαφές μας με τους σκιώδεις υπήρξε μια συμβιβαστική διάθεση από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε με αποτελεσματικό τρόπο και με μεγάλη ταχύτητα, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο. Το πρώτο που θα ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι είμαι έμπλεος αισιοδοξία πλέον σχετικά με, τον δυνατό, με τη δυνατότητα σεβασμού του χρονοδιαγράμματος. Η ψηφοφορία εδώ λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή θα γίνει το Φεβρουάριο και νομίζω ότι θα καταλήξουμε στην Ολομέλεια τον μήνα Απρίλιο. Να υπογραμμίσω κάτι επιπλέον ότι αυτό στάθηκε εφικτό γιατί υπήρξε μια μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στα διάφορα κόμματα και τις πολιτικές ομάδες οι οποίες ε, εδώ αντιπροσωπεύονται σχετικά με την δυνατότητα ε, προστασίας του καταναλωτή. Αυτό ήταν το βασικό θα έλεγα πεδίο εργασίας μας. Ένα άλλο θέμα στο οποίο έχουμε επιμείνει ιδιαίτερα είναι η λεγόμενη λογική απροποίηση. Προσπαθήσαμε εμείς να απλοστεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την οδηγία αυτή έτσι ώστε να μην χρειαστεί σύντομα να επανέλθουμε στην επανεξέτασή της. Έχει υποθεί άλλωστε επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε μέσα από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε ε, τις ε, δυνατότητες τις νέες οι οποίες υπάρχουν περνώντας από το PS1 στο PS2 δεν αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα ιδιαίτερα δεν αλλάζει το λεγόμενο νομικό πλαίσιο αλλά υπάρχει μία προσαρμογή θα έλεγα Θέλουμε το νέο διακανονιστικό πλαίσιο να εξυγχρονιστεί και να γίνει ε, πιο ε, κατανοητό. Βλέπουμε λοιπόν τι νέες πραγματικότητες έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε ε, και τι κάνουμε για να το πετύχουμε. Σαν παράδειγμα ασφάλεια, εγγύηση της ασφάλειας των συναλλαγών, αποτροπή των απατών και επίσης ε, δυνατότητα σεβασμού των ε, βασικών αρχών που διέπουν ε, την συγκέντρωση των τραπεζικών δεδομένων. Όλα αυτά τα κάναμε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να κλείσω εδώ λέγοντας αυτό το οποίο είπα στην αρχή. Είμαι αισιόδοξο. Ελπίζω να συνεχιστούν οι εργασίες μας με μεγάλη ταχύτητα και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλους τους σκιώδεις, όλους τους βοηθούς του, τους συνεργάτες του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα έγιναν με ε, τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στον Πάμπλο για το επόμενο θέμα, τις προμήθειες για τις ε, συναλλαγές με κάρτες θα ήθελα να ξεκινήσω εκεί που σταμάτησε ουσιαστικά ο συνάδελφος και φίλος Φεϊό. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω λοιπόν και τους συνεργάτες μου και τους συνεργάτες των σκιωδών εισηγητών και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια της έκθεσης αυτής προσπαθήσαμε να καθορίσουμε τέσσερις προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η διαφάνεια, η συγκέντρωση στις στο σεβασμό των αρχών της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς. Por último, y no menos importante, la Και φυσικά κυρίως να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Οι προτεραιότητες αυτές είναι δύσκολο να τις εξισορροπήσει κανείς. Μερικές φορές τα συμφέροντα είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να εξισορροπήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτές τις τέσσερις πρωτοβουλίες. Κάποιοι κάνουν κριτική λέγοντας ότι το ανώτατα όρια, η θέση ορίων στις προμήθειες θα επηρεάσει αρνητικά τα άλλα κόστη που συνδέονται με μια πιστοτική κάρτα. Ε, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Κανένας δεν αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο. Αλλά στη χειρότερη περίπτωση, ε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο τη διαφάνεια και θα έχουμε πετύχει τη διαφάνεια. Γιατί όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί την πιστοτική του κάρτα, θα γνωρίζει επακριβέστατα το τι ακριβώς καλείται να πληρώσει. Τώρα έρχομαι στις τροπολογίες. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τις τροπολογίες και για τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στην έκθεση στην οποία είμαι. Καταρχάς το ενιαίο το μοναδικό άρθρο σχετικά με το πεδίο εφαρμογής. Όπως όλοι γνωρίζετε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει τα συστήματα τα οποία αποτελούν τμήμα της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τα ανώτατα όρια των προμηθειών και τις προβλέψεις του άρθρου 7 σχετικά με το διαχωρισμό των πιστοτικών καρτών και των ε, κέντρων επεξεργασίας. Ε, αυτά είναι θέματα τα οποία συζητάμε με τους συζητητές ακόμα. Ένα θέμα όμως ε, τίθεται. Υπάρχει μια δυσκολία με, με, τα, με τις προμήθειες των λεγόμενων τριμερών συστημάτων. είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλουμε ένα όριο σε σχέση με αυτό. Σχετικά με το άρθρο 2 στους ορισμούς, εδώ ε, πιστεύω ότι καταλήγουμε με τους σκιώδεις σε μια κάποια συμβιβαστική λύση σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι είναι μια πιστοτική κάρτα και τι είναι μια χρεωστική κάρτα για τα ΚΑΠ τώρα, όπως επίσης και για την περίοδο εφαρμογής ε, ε, των άρθρων 3 και 4. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει συνένεση ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα το ανώτατο όριο το 0,3. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες διαφορές και υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τα ανώτατα όρια των ε, συναλλαγών με πιστοτικές κάρτες η συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή και ελπίζω να καταλήξουμε, να αναζητήσουμε και να καταλήξουμε στην πιο καλή συμβιβαστική λύση. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να επιμείνω λέγοντας ότι η συζήτηση θα πρέπει να λάβει υπόψη να ακριβώς το τι συνέπειες θα έχει η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων για τις πιστοτικές κάρτες στις διάφορες χώρες. Υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει ε, τις πληροφορίες περισσότερες ε, για τα θέματα αυτά. Σχετικά τώρα με το άρθρο 8 και de la Comisión λεγόμενη, το, το, το co-budgeting. Η αδυναμία να έχει ένας χρήστης ε, ένα μέσο πληρωμών προεπιλεγμένο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και ότι θα πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό αν θέλετε τέτοιο μέσο είναι ένα, μια περιπλοκότητα περιττή, μια επιπλέον δυσκολία κατά τη στιγμή της πληρωμής και μια αιτία καθυστέρησης. Θα ήθελα να υπάρξει μια συμβινένεση εδώ ένα συμβιβασμός έτσι ώστε πράγματι να υπάρχει η δυνατότητα προεπιλογής από ο πλευράς του καταναλωτή ενός ή περισσότερων εμπορικών σημάτων και όχι κάθε φορά που κάνει μία πληρωμή να επιλέγει κάθε φορά ακριβώς το σήμα Νομίζω λοιπόν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα, αν το επιθυμεί ο χρήστης, να προεπιλέξει το εμπορικό σήμα ή το σύστημα ε, πληρωμών το οποίο, επιλογεί, το οποίο επιλέγει για να κάνει την ε, συναλλαγή του. Σχετικά τώρα με το άρθρο 10 για τη δυνατότητα αποδοχής όλων των καρτών το λεγόμενο Common All Card Rule. Έχω την αίσθηση και εδώ σκέφτομαι σαν καταναλωτής ότι θα πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση των κανόνων υποχρεωτικής αποδοχής πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει έτσι ώστε η πιστοτική μας κάρτα να μπορεί να γίνεται δεκτή ε, σε ένα εμπορικό ε, ταμείο κτλ. Αν τώρα ένας έμπορος επιλέγει το ποιες θα χρησιμοποιεί ή όχι, αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους χρήστες και θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο έχουμε στο νου μας, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή περισσότερο τις πιστοτικές κάρτες και με μεγαλύτερη ταχύτητα και το να μην στην περίπτωση που δεν δέχεται μία, μία πιστοτική κάρτα τότε θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση είτε μετρητής είτε κάτι άλλο και ό,τι άλλο χρειάζεται απαραίτητο. Είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα της συμβιβαστικής λύσης την οποία αναζητούμε στα πλαίσια του άρθρου 10 θα πρέπει να είναι συμβατό με την έκθεση και του συναδέλφου Φεγιό partidario de que se elimine la posibilidad eh, η δυνατότητα ενός εμπόρου να απορρίψει μια πιστοτική κάρτα υπάρχει, αλλά πρέπει να επιτρέπουμε ταυτόχρονα στους ε, εμπόρους ίσως να βάζουν ένα επιπλέον τέλος λόγω ακριβώς του υποχρεωτικού αποδοχής ε, όλων των πιστοτικών καρτών. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές γραμμές. Εγώ θα ήθελα να ακολουθήσουν αυτές τις κατευθύνσεις ε, οι προτάσεις μου, αλλά είμαι στη διάθεσή σας και θα λάβω υπόψη ε, ότι σας απασχολεί. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πρώτος και των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω με τις συνήθεις ευχαριστίες προς τον εισηγητή. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που για μας είναι δύσκολα και θα ήθελα να βρούμε από αυτόν κάποιο συμβιβασμό. Λοιπόν, βασίζομαι στο εξής. Χρειαζόμαστε μια σαφή προοπτική συνεπή για την εσωτερική αγορά. Υπάρχει κατανομή στα 28 κράτη-μέλη και υπάρχουν και θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και κινητικότητας διαμεθοριακής. Υπάρχουν περιορισμοί, αλλά πρέπει να σεβόμαστε πάντοτε το στόχο της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν μερικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να συμφωνήσουμε και θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το σημαντικότερο τμήμα της πρότασης της Κομισιόν, την διαχείριση από τρίτους. Μέσω της χρήσης όμως κοινών κανόνων. Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό υπόδειγμα ή πρότυπο που έχουμε. Δεν χρειάζονται αναγκαστικά κάθε φορά συμφωνίες και συμβόλαια με προμηθευτές ή άλλους τρίτους αλλά κοινοί κανόνες και πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταλαβαίνουν τι ακριβώς ισχύει. Οι διαδικασίες να ελέγχονται πιο φανερά από ό,τι μέχρι τώρα και ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι έχει ασφάλεια η δοσοληψία του. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να συνεργαστούν για να αποσαφινιστούν τα πάντα. Η συζήτηση μέχρι τώρα ήταν επικοδομητική, αλλά πρέπει να προσέξουμε να βρούμε μια λύση η οποία να λειτουργήσει με πραγματικούς όρους. Επίσης σημαντικό είναι η εισφορά που πληρώνουμε να μην είναι, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά. Καμιά φορά σημειώνονται προβλήματα γιατί οι εισφορές ε, πληρώνουν ε, δαπάνες που δεν πρέπει να τις φέρει ο καταναλωτής. Πρέπει να έχει αντίθετα την εντύπωση ότι όλα είναι εξισορροπημένα και δίκαια. Στις χώρες μέλη καμιά φορά απαγορεύονται τέτοιου είδους εισφορές επιβεβαρημένες. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεπή εσωτερική και λογική εσωτερική αγορά, θεωρώ ότι πρέπει η πρόσθετη αυτή εισφορά που επιβαρύνει κυρίως τους τρίτους, που για να πληρωθούν οι τρίτοι μάλλον, είναι κάτι που θα μπορούσε να περιοριστεί. Εδώ η θέση της Κομισιόν είναι επαρκής να σκεφτεί την περίπτωση της απαγόρευσης αυτής της βεβαρημένης εισφοράς. Θα ήταν αυτό πιο καλό για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Καφέ Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε αν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση για τις ε, πρόσθετες αυτές τις φορές. Εγώ είμαι ανοιχτός και θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω διάφορες τεχνικές εναλλακτικές λύσεις. Καταλήγω λέγοντας το εξής. Γενικώ πρέπει να ενδυναμώσουμε την προστασία του καταναλωτή και σε αυτό το θέμα η πρόταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλντίνη, αλλά δεν είναι παρόν. Η κυρία Σόφη Ιντβέλτ ή κάποιος που να την αντικαθιστά. Νίλς, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστώ για αυτή την ισορροπημένη έκθεση την οποία και στηρίζω σε μεγάλο βαθμό. Έχω βέβαια καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ε, της ε, προμήθειας τόσο για τις πιστοτικές όσο και για τις χρεωστικές κάρτες. Και εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο ανώτατο όριο θα είναι τροχοπέδι και πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να είναι αυτού του ύψους ώστε να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος ε, των συναλλαγών. Στη Σουηδία αλλά και στη Φινλανδία οι κάρτες είναι ευρέως ε, δεδομένες. Στο Ελσίνκι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την ψωτική του κάρτα για να αγοράσει και εισιτήριο στο λεωφορείο ή ένα καφέ σε ένα μικρό καφενείο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όμως αν τελικά αυτές οι συναλλαγές ρυθμίζονται με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προκαλούν ζημιά στις τράπεζες οι τράπεζες δεν θα προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στους ε, μαγαζάτορες και έτσι θα καταστεί απαραίτητο να έχει κανείς ε, περισσότερα χρήματα μετρητά ε, πάνω του. Αυτό όμως δεν ξέρουμε αν ε, εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες ε, καταστημάτων. Αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν ε, καινοτομίε, να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες με ταχύτητα. Βεβαίως αν συμβεί κάτι τέτοιο οι τράπεζες δεν θα έχουν κανένα κίνητρο να δημιουργήσουν ένα σύστημα απαραίτητο, δηλαδή να γίνονται συναλλαγές κάτω από 28 ευρώ, οι οποίες όμως θα είναι ζημιογόνες. Οι πληροφορίες μας λένε ότι για κάθε συναλλαγή, η κάθε συναλλαγή κοστίζει 45 cent, άρα δηλαδή μία συναλλαγή γύρω στα 20 ευρώ αξίζει τον κόπο εάν ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το 60% όπως σας είπα των συναλλαγών στη Σουηδία και τη Φιλανδία είναι με κάρτες αλλά κάτω από 20 ευρώ. Άρα αν υπάρχει αυτό το ανώτατο όριο τότε οι ε, κατέχοντες ιδιοκτήτες καρτών ε, θα τιμωρούνται και θα προκύπτει και ζημιά που όπως σας είπα θα ανέρχεται σε περίπου 0,9% του συνόλου του ποσού. Εάν λοιπόν όπως σας είπα το ανώτατο όριο εισαχθεί για το ανώτατο κόστος, θα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο για το κατώτατο κόστος ε, της ε, συναλλαγής. Εγώ προσωπικά προτείνω ε, να υπάρχει ένας ε, μέσος όρος, σταθμισμένος μέσος όρος. Και είμαι και υπέρ της ε, διαφάνειας. Βέβαια, αν οι εθνικές εποπτικές και τραπεζικές αρχές επιβάλλουν κάποιες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, τότε καταλαβαίνω ότι θα προκύψουν προβλήματα. Η δεύτερη πρόταση είναι σχετικά με το όριο για τις πιστοτικές κάρτες. Εγώ προτείνω να διαγραφεί το όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους χρήστες όλων των καρτών. Η τρίτη παρατήρηση αφορά τον ορισμό συναλλαγής με χρεωστική κάρτα. Μετά από 48 ώρες ε, η ε, το ποσό χρεώνεται και αυτό είναι ένα κίνητρο για τις τράπεζες να καθυστερήσουν τη συναλλαγή για δύο περίπου ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να επανέλθουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τέλος θέλω να πω ότι είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει δώσει μια αξιολόγηση επιπτώσεων για το τι ε, συνέπειες θα προκύψουν στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί όπως είπα και στην αρχή, σε ορισμένα κράτη-μέλη οι κάρτες είναι ευρέως διαδεδομένε σε άλλα πάλι όχι. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Τώρα, αν αντικαταθιστάτε κάποιον σκιώδη πρέπει να ακολουθείτε τη γραμμή του σκιώδους ενώ εσείς δεν ακολουθήσατε τη γραμμή του σκιώδους που, που αντικαθιστούσατε είχατε δική σας γραμμή Νομίζω πρέπει να το αποσαφηνίσω αυτό. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές απόψεων και ο Νίλς αποσαφήνισε ότι μιλάει για τις δικές του τροπολογίες. Εντάξει, θεμητό. Αλλά πρέπει να αποσαφηνίσω ότι δεν ήταν λόγος εξ ονόματος της Σόφη. Ο κύριος Μπαλντίνη τώρα. Μα τι πρόβλημα έχει εκεί κάτω. Κοιτάξτε, πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο Νίλς. Ε, Πώς μπορεί να το κάνει ο Νίλης ε, τη στιγμή που από τη δική του την πολιτική ομάδα το ποσοστό είναι μεταξύ 0,1 και 0,4 και η κυρία Ιντφέλτ έχει προτείνει 0,1 εκ μέρου των φιλελευθέρων. Πώς μπορεί να συμβιεστεί αυτό, να προτείνουμε το μέσο όρο 0,3? Κοιτάξτε, αν θέλετε να μετράτε πόντου σε πολιτικέ ομάδε, εμένα δεν με νοιάζει, κάντε το. Εγώ θέλω απλά να επικρατεί τάξη, πρώτα να μιλάνε και ο και μετά ένα επίσημο εκπρόσωπο. Ε, θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλντίνη, γιατί έχει έλθει μεταξύ ο κύριο Μπαλντίνη στην αίθουσα. Παρακαλώ κύριε Μπαλντίνη. Ευχαριστώ. Ε, θα μιλήσω κροατικά αφού υπάρχει και η διερμηνία. Λοιπόν, πρώτον, για την πρόταση της Κομισιόν ως προς το θέμα των συναλλαγών και των ποσών που παίρνουν για αμοιβή οι οργανισμοί πιστοτικών καρτών. Είναι πολύ εξαιρετική πρόταση για διάφορους λόγους. Ένας από τους οποίους είναι ότι δίνεται έτσι η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν κάποια διαφάνεια στις δοσοληψίες τους με τις πιστοτικές κάρτες. Τώρα θα μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν πόσα πληρώνουν για την κάρτα τους. Και όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, πράγματι Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά αυτό το ξέραμε. Έχουμε λάβει έγγραφα της Κομισιόν που μας έδειχναν τι χάσμα υπάρχει στα ποσοστά που παίρνουν οι τράπεζες σε σύγκριση με άλλες μορφές πληρωμών. Στη Μεσόγειο είναι περίπου 30% και στη Βόρεια Ευρώπη, βορειοδυτική συγκεκριμένα, Μέχρι 70%. 70% όλων των πληρωμών γίνονται με κάρτες. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό διότι μας δίνει μια ιδέα των διαφορών που υπάρχουν στο ρυθμό χρήσης της πιστοτικής κάρτας στην Ένωση. Δεν αφορά όμως μόνο τον όγκο των δοσοληψιών το θέμα. Εδώ μιλάμε και για τα, την προμήθεια των τραπεζών. Και εδώ η πρόταση της Κομισιόν δεν στοχεύει μόνο σε μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και στην ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της κάρτας. Αυτό είναι στο κάτω-κάτω και ο στόχος της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν ολόκληρης. Δεν είναι τίποτα καινούριο είναι καλό που μπορούμε να το συζητήσουμε. Ακούσαμε εξαιρετικές προτάσεις του κυρίου Ζάλμπα. Και εξ ονόματος της ομάδας μου, ως σκιώδης δηλαδή, μπορώ να πω ότι καταθέσαμε προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της πρότασης της Κομισιόν ακόμη περισσότερο. Είναι ήδη καλή όπως σας είπα και αναφέρεται στα βασικά θέματα και προβλήματα, θέλει να ενοποιηθεί το σύστημα των δοσοληψιών με κάρτα, να μειωθούν οι προμήθειες των ραπεζών για να είναι πιο, και να γίνει πιο εύκολο για τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις πιστοτικές κάρτες πληρώνοντας λιγότερα λιγότερη προμήθεια αλλά πρέπει να η διαδικασία να είναι διαφανής έχουν το δικαίωμα οι πολίτες μας να γνωρίζουν πόσο τους κοστίζει η χρήση της πιστοτικής τους κάρτας πόσα παίρνει η τράπεζα, γιατί ποσοστά μιλάμε. Ακούσαμε, την πρότα... ξέρουμε την πρόταση της Κομισιόν στη Γερμανία, περίπου 1,8, στη Δανία 1,1 και 0,1 και υπάρχουν και όλα τα ενδιάμεσα ποσά. Αν τώρα καταλήξουμε σε μέσο όρο 1,2 πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Δανία έχει χαμηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο. Αλλά οι Δανείοι πληρώνουν 80% βέβαια των δοσοληψιών τους με πιστοτική κάρτα. Άρα η ενοποίηση της αγοράς θα αυξήσει την διαφάνεια και τον όγκο των δοσοληψιών με πιστοτικές κάρτες. Και έτσι θα μπορεί να αποδυναμωθούν ορισμένοι δομεί της οικονομία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις προτάσεις του κυρίου Σάλμπα. Κάνω και εγώ ότι μπορώ να βοηθήσω με την ομάδα μου για να βοηθηθούν, υποβοηθηθούν όλα αυτά και να πετύχουμε όσο περισσότερα μπορούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα σε έναν από τους πρασίνους. Δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο για τις υπηρεσίες πληρωμών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εισαγωγικά και εντάχει. Έχω την αίσθηση και η πολιτική μου ομάδα ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο μαζί με τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές για να πετύχουμε τον διπλό στόχο αυτής της οδηγίας από τη μία δηλαδή να βελτιωθεί ο ανισμός, να είναι πιο δίκαιος και πιο ασφαλής, διεύρυνση του πεδίου των συστημάτων πληρωμών, προς τον συμφέρον ταυτόχρονα των καταναλωτών. Δεν θα παρουσιάσω τον κατάλογο των συμφωνιών μας μετά από τις συμβιβαστικές προτάσεις των εισηγητών. Είναι πολλές και τα έχουμε πει. Θα πάρω όμω δύο παραδείγματα επιφυλάξεων που έχουμε και να κάνω και δύο σκέψεις ε, ίσως λίγο γενικότερες επί της ουσίας πάντα. Δύο παραδείγματα επιφυλάξεων που μας διακατέχουν. Πρώτον, το όριο των λεγόμενων βοηθητικού τύπου συναλλαγών, όπως ας πούμε ε, οι ήχοι των κινητών τηλεφώνων που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1 της παραγράφου 3 θα πρέπει να τύχουν ενός του ορίου και τα κράτη-μέλη θα μπορούν και ενθαρρύνονται συγγνώμη, να τη Τώρα για την υποχρέωση διατήρησης των στοιχείων είμαστε υπέρ των συμβιβαστικών προτάσεων των εισηγητών εκτός από ένα σημείο την δυνατότητα για τις εθνικές υπηρεσίες να αποκλίνουν των συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως παρουσιάζεται και προτείνεται στην 2β. Υπάρχουν δύο επιπλέον κομβικά σημεία τα οποία δεν έχουν τύχει αντιμετώπισης από τις συμβιβαστικές προτάσεις. Πρώτον, το θέμα της πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών και δεύτερον η νομική ευθύνη στην περίπτωση δημοσίευσης των ατομικών στοιχείων σε έναν παροχέα υπηρεσιών πληρωμών, έτσι όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 66. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της υπερβολικής τιμολόγησης, της υπερτιμολόγησης. Έχουμε μιλήσει με την Επιτροπή για το θέμα αυτό και μας διαφώτισε αρκετά. Υπάρχει το θέμα στο άρθρο 55 των υπερβολικών τελών και εδώ συνεχίζουμε να προτείνουμε μια πλήρη και απόλυτη απαγόρευση αυτού του συστήματος υπερτιμολόγησης. Ένα σύστημα το οποίο σε ορισμένες χώρες λειτουργεί χωρίς να υπάρχει. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους ο Μπάς τώρα. Κοιτάξτε, ομιλώ και εγώ εκ μέρους των ε, πρασίνων και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχήν, Μιλάμε για τι διατραπεζικέ προμήθειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίω γιατί μιλάμε για την προστασία του καταναλωτή. Και έτσι καλωσορίζουμε την πρόταση τη ε, Κομισιόν, ε, συζητώντα για του ε, συμβασμού. Θέλουμε να παραμείνουμε κοντά στην πρόταση της Επιτροπής, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν επιτύχει τη σωστή ισορροπία. Βεβαίω, Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να επιτύχουμε συμβασμό. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή που το κατάφερε αυτό. Ε, θέλω να πω το εξή, ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το άρθρο 3-4, εκεί όπου αναφέρονται τα διάφορα επίπεδα ανώτατων ορίων. Νομίζω, όπως είπε και ο εισηγητής, ε, μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε σε αυτά τα ανώτατα όρια για τις ε, πιστοτικές κάρτες. Για τις χρεωστικές ορίζουν τώρα και ένα καθαρό επίπεδο, όχι μόνο την αναλογία που θα μπορούσε να είναι τα 7 cent. Γιατί αν σκεφτείτε πολύ μικρά ποσά για τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μια χρεωστική ε, κάρτα, ας πούμε 10 ε, ευρώ, τα 7 cent είναι πάρα πολλά. Ίσως λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε ε, το ανώτατο όριο και όχι να είναι 7, να είναι λίγο πιο κάτω. Ε, στη Δανία ε, είναι 0, στο Βέλγιο 5 cent και εμείς είμαστε υπέρ του μηδενικού, της μηδενικής χρέωσης, αλλά για να υπάρξει συμβασμός, εντάξει μπορούμε να συζητήσουμε. Χαμηλότερο πάντως επίπεδο, καλό είναι ότι προβλέπεται ένα σαφές ε, προκαθορισμένο όριο για τις ε, χρεωστικές κάρτες. Κατόπιν, τη θέση σε ισχύ. Εμείς θέλουμε ε, να το συζητήσουμε αυτό με την Επιτροπή και η Επιτροπή κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε θέση σε ισχύ διασυνοριακά και σε εσωτερικό επίπεδο. Εμείς θέλουμε ενδεχομένως να υπάρξει ένα και μόνο άρθρο που να αφορά γενικά τη θέση σε ισχύ. Εφόσον όμως τώρα συζητάμε για θέση σε ισχύ και μιλάμε για ένα χρόνο, Άρα δηλαδή αυτό είναι πολύ μακριά από αυτό που προτείνει η Κομισιόν για τη διασυνοριακή θέση σε ισχύ. Πρέπει αυτό να το συζητήσουμε ισκιώδης, αλλά ε, θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Επιτροπής επί του θέματος. Κατόπιν, όσον αφορά το άρθρο 8 το περίφημο co-budgeting, όπως το είπε και ο εισηγητής. Νομίζω κατέστη σαφές στη συνεδρίαση των σκιωδών ότι για μας δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ε, αλλάξουμε αυτό το co-budgeting που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μία από τις ε, μεγάλες συζητήσεις που θα έχουμε είναι για το άρθρο 10 Εκεί θέλω να εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν θέλουμε να αποκλίνουμε από την πρόταση Επιτροπής και θεωρούμε ότι με αυτές τις κάρτες, αν εγκατασταθούν, ε, θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι καταναλωτές στις κάρτες γενικότερα. Αυτό που εμάς μας ανησυχεί είναι ότι αν τελικά χρησιμοποιηθούν αυτές οι κάρτες, όσοι είναι υπέρ των χαμηλών εισφορών θα αναγκαστούν να πληρώνουν τελικά υψηλές εισφορές, γιατί όλοι έχουν ας πούμε μία βίζα. Για μας είναι πολύ σημαντικό στο λιανικό εμπόριο να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να απορρίψει μία κάρτα. Εμείς ε, στηρίζουμε της δυνάμεις αγοράς στην περίπτωση αυτών των καρτών. Γι' αυτό λοιπόν στο άρθρο 10 θα θέλαμε να παραμείνουμε κοντά στην πρόταση της ε, Κομισιόν. Και εκεί δεν συμφωνούμε με τον εισηγητή. Επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό συζητήθηκε στην συνάντηση των σκιωδών, ο σκιώδης των φιλελευθέρων έκανε μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε να υπάρχουν νέες προτάσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τους σκιώδης ηγητές και μετά θα δούμε τι θα γίνει με την ε, ψηφοφορία. Αυτές είναι οι σημαντικές μας προτάσεις. Νομίζω ότι τώρα τα πάμε πάρα πολύ καλά και νομίζω αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον και για το άρθρο υπαριθμών 10. Σας ευχαριστώ πολύ. Άσυλο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας μου. Και για τα δύο θέματα, για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ τον Διέγκο και τον Πάμπλο Καταρχήν να σχολιάσω μερικά για την οδηγία πληρωμών 2, για τις ψηφιακές εξαιρέσεις. Ο λόγος που θέλησαμε να καταθέσουμε τροπολογίες στο 3.1 ήταν για να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες. Εμείς δεχόμαστε ότι ο συμβιβασμός του κυρίου Φέο πρέπει να, να αρκέσει σε όλους, να αποκλειστούν δηλαδή οι φιλανθρωπικές δαπάνες. Ζητώ όμως από την Κομισιόν Ερωτώ την Κομισιόν, τη ζητώ να σχολιάσει, υπάρχει νομική σαφήνεια για αυτή τη συμβιβαστική πρόταση. Για τα TPP τώρα. Οι American Express και οι Diners πρέπει να εξαιρεθούν και αυτές διότι λειτουργούν με διαφορετικό ε, πρότυπο λειτουργικό από ότι με Κίνα που λειτουργούν με τετραμερή κατανομή. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να εμποδιστεί η διμερή συνεννόηση των παραγόντων αυτών με τους εμπόρους. Εξάλλου πολλοί έμποροι δεν δέχονται αυτές τις κάρτες γιατί τους κοστίζουν πιο πολύ. Και εδώ υπάρχει η σχέση της οδηγίας με τον μύθο. Υπάρχει όντως ελευθερία, κανείς δεν εμποδίζει τον έμπορο να απορρίψει μια κάρτα. Τώρα για τα δίκτυα και την οδηγία ασφάλειας των πληροφοριών. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη όλα αυτά, ούτε ξέρουμε τελικά ποιες θα είναι οι προτάσεις και γι' αυτό να αναφερθούμε σε αυτό το σχέδιο οδηγίας στο PSD2 μου φαίνεται ότι δεν είναι σωστό. Οι υποχρεώσεις του PSP υπό το NIS δεν είναι σαφής και συγκρίσιμα μέτρα που προβλέπει ήδη το κείμενο της PSD2 είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να μην αναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα η οδηγία μυφ. Καταρχήν ο συμβιβασμός για τις χρεωστικές κάρτες. Ο συμβιβασμός με το 2% δεν γίνεται δεκτός από την ομάδα μου, αλλά δεν έχουμε πιστεί από το 0,3% για τις πιστοτικές κάρτες. Εμείς πιστεύουμε ότι αν βάλουμε τόσο χαμηλά το όριο θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Νομίζουμε ότι θα βλαφτεί ο ανταγωνισμός. Δηλαδή οι μικρότερες πιστοτικές εταιρείες, εταιρείες πιστοτικών καρτών δεν θα μπορούν πια να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες και μπορεί να σταματήσουν και τη λειτουργία τους. Νομίζω ότι η Κομισιόν δεν έχει λάβει υπόψη της το γεγονός ότι δεν βγάζουν πιστοτικές κάρτες μόνο τράπεζες και η τέτοια, μια τέτοια μείωση των προμηθειών τους που στη χώρα μου θα αντιπροσώπευε το 0,85% θα κατέληγε μάλλον σε επιβολή ετησίων εισφορών για τον κάθε χρήστη. Πράγμα το οποίο δεν θέλουν να το πληρώσουν οι πελάτες τους. Τώρα για τις διάφορες άρες επιβαστικές προτάσεις. Είμαι υπέρ του κυρίου Λάγκεν 176 που μιλάει για 0,8% στην αρχή που θα μειωθεί σε 5 χρόνια σε 0,3%. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό συμβιβασμό και η ομάδα μου θα μπορούσε να τον υποστηρίξει εάν και ο εισηγητή το δέχονταν. Νομίζω ότι η, αναμονή, διετής αναμονή όμως είναι υπερβολική και οι σκιώδεις γενικά θεωρούν ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορούσε να γίνει η αλλαγή αυτή. Όσο για το χωρισμό scheme και processing. Υποστηρίζω την πρόταση του κυρίου Ζάλμπα. Αν είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία πιστοτικών καρτών να διαχειρίζεται μόνη της όλες τις δοσοληψίες μπορεί αυτό να την επιβαρύνει πολύ. Το πρόσθετο κόστος για τη χρησιμοποίηση τρίτου θα το επιβαρύνουν, θα επι... πληρωθεί και από τους καταναλωτές και από την εταιρεία. Γενικά δεχόμαστε τις προτάσεις του κυρίου Ζάλμπα. For the GUI, uh, Ja, danke, Sharon. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ε, είμαι αρμόδιος ως Σκιώδης και για τις ε, δύο εκτέσεις. Επειδή χτες είπες ότι είσαι μαρξιστής, το είπες για τον εαυτό σου, πολύ ευχαριστώ. να έρθεις και εσύ αν θέλεις. Δυστυχώς γίνονται και άλλα σχόλια εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την μέχρι τώρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και κατά τη δική μας άποψη η πρόταση της Επιτροπής είναι μια καλή πρόταση, αναμφισβήτητα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήδη έχουν λεχθεί πολλά, πολλά εξ αυτών τα υποστηρίζω, γι' αυτό θα περιστώ σε λίγα μόνο θέματα τα οποία ε, με απασχολούν περισσότερο ως καταναλωτή σχετικά με το ΜΥΦ. Θέλω να πω, όχι ΜΥΦΙΤ, άλλο το ΜΥΦΙΤ, εγώ μιλάω για το ΜΥΦ. Θέλω να υπογραμμίσω ότι κατά την άποψή μας το co-budging ε, έχει νόημα. Ε, η αιτιολογία είναι γνωστή ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τον ε, καταναλωτή να δουλεύει με μία κάρτα από το να έχει πολλά προγράμματα στη διάθεσή του. Κατά την άποψή μας ε, όταν υπάρχουν πολλές κάρτες δημιουργείται ανταγωνισμός. Βεβαίως ε, αυτό από την άλλη σημαίνει ότι ε, μειώνεται το κόστος. Τις δύο βασικές μου παρατηρήσεις θέλω να τις κάνω για την οδηγία, την PSD. Υπάρχουν δύο θέματα που για τον καταναλωτή είναι πολύ σημαντικά. Έχουν γίνει κάποια βήματα στη σωστή κατεύθυνση, Θέλω όμως να επισημάνω ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Υπάρχει το πρόβλημα με τα TPP, τους Party Providers, όπου τα τραπεζικά δεδομένα μέχρι τώρα μεταβιβάζονται σε ένα τρίτο μέρος μαζί με το PIN και πολλά άλλα στοιχεία για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό όμως ε, κατ' ουσία σημαίνει ότι ο καταναλωτής, ο πελάτης ε, πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία που τον αφορούν για να μπορεί να πληρωθεί από ένα τρίτο μέρος. Mm. Αυτό όμως συνεπάγεται πολλούς κινδύνους. Και μόνο αυτό αλλά όταν μεταβιβάζονται τραπεζικά δεδομένα, ε, πολλές φορές ε, ε, για λόγους για αμέλειας μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα και μετά αν κανείς κατηγορηθεί για αμέλεια καταλαβαίνετε ότι δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Οι ασφάλειες πλέον δεν καλύπτουν σε περίπτωση απώλειας τον αριθμό του ΠΙΝ, δηλαδή την πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει κανείς να τον διαχωρίζει, να έχει ένα πιν για γενικότερη πρόσβαση και ένα άλλο πιν που θα αφορά μόνο τις πληρωμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας το έχουν επισημάνει οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτή. Και γι' αυτό το λέω και εγώ, για να πω ότι είναι μια πρακτική λύση που θεωρώ ότι είναι και σημαντική και τη στηρίζω και λέω να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε ήδη με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ε, έγινε λόγος και για αριθμό ΤΑΝ και αυτό είναι μια λύση. Μετά, από πλευράς του καταναλωτή, τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία, υπάρχει εξή ε, πρακτική. Μέσα σε δύο μήνες μπορεί κανείς ε, να ανακαλέσει ποσά. Αυτό βέβαια σπάνια γίνεται και κατόπιν τούτου όλο αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο. Δεν υπάρχει κίνδυνος ε, κατάχρησης. Όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές. Θέλουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα και να νιώθουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή τι θέλει κανείς, αν αισθανθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα με το συνεργάτη του και του είχε βάσει κάποια χρήματα, να μπορεί να τα ανακαλέσει, να τα πάρει πίσω. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει τον πελάτη να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτή τη ε, διαδικασία πληρωμών. Η δυνατότητα ανάκλησης ποσών να προβλέπεται στην οδηγία. Αν βέβαια αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια ενός κράτους μέλους, τότε κατά τη γνώμη μου υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, οι επιχειρηματίες από τη Γερμανία, όπου θα συνεχίσουν να μπορούν να ανακαλούν ποσά, πάνε σε μια άλλη χώρα. Εκεί όμως δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης ποσού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δημιουργείται αδιαφάνεια, δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή να αγοράζει κανείς κάτι σε μια χώρα και να μην ξέρει έχει τη δυνατότητα ανάκλησης ή όχι. Ποιες διατάξεις ισχύουν, οι γερμανικές, οι γαλλικές, κάποιες άλλες. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να επιδιώξουμε σαφήνεια, να αναζητήσουμε μια λύση η οποία θα ισχύει για το σύνολο της κοινή αγοράς και όχι για μεμονωμένα κρατημέλη. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα να κάνω και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από το EFD. Έχω αρκετούς εδώ ομιλητές. Αν θα μιλήσει η Επιτροπή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητά σας. Λάγκεν, Γκοζές, Σμιτ, Κλίντς όταν επιστρέψει, αν επιστρέψει και Τάισεν. Βένα. Fox έχει ja äh, einen meiner Änderungsanträge schon ο συνάδελφος Φόξ αναφέρθηκε ήδη σε μία από τις ε, τροπολογίες μου. Ανάλογα ή θα είναι το 0,7% ή το 0,8% ε, θα προβλέπεται αυτό το ποσοστό για πέντε χρόνια και όχι για μία συγκεκριμένη μέρα. Ξέρετε, αυτό το μοντέλο ε, αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένο στα τέλη περιαγωγής. Ε, σιγά σιγά τα μειώσαμε και έτσι κατορθώσαμε να προάγουμε και τον ανταγωνισμό και οδυνηρές συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω αυτές οι δικές μου τροπολογίες, οι δύο, είναι πολύ καλές, ισχύουν, μπορούν να εφαρμοστούν για τα θέματα που συζητάμε και όλες οι άλλες ε, τροπολογίες της κυρίας Ιντφελτ το 0,0 ή της κυρίας Βόρτμαν Κόλ, αυτές δεν πρέπει να τις συμπεριλάβουμε σε συμβαστική πρόταση, γιατί τις θεωρώ ουτοπικές και κάποιος στη τελική ανάλυση πρέπει να πληρώσει. Το πιο δίκαιο είναι ο ανταγωνισμός να γίνεται ανάμεσα στις κάρτες και να υπάρχει μια διαφάνεια όχι όμως ε, εμείς με τις προτάσεις μας να δημιουργούμε αδιαφάνεια. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος μας. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα συμβαστική πρόταση για τα συστήματα τριών ή τεσσάρων μερών. Εγώ πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε ε, τον θεμητό ανταγωνισμό μέσω των δικών μας των ρυθμίσεων, των εξαιρέσεων ή των ε, κατώτατων ή ανώτατων ορίων να είναι το 5% της αγοράς παραδείγματος χάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ να μην οδηγήσουμε με τον τρόπο αυτό στο να προτιμάει ο καταναλωτής όπως και επιχειρήσεις αμερικανικά συστήματα. Ίσως ε, αυτό να είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που να απασχολεί το City του Λονδίνου. Δεν μπορούμε όμως εμείς να αποφασίζουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα καλό συμβιβασμό ε, και γι' αυτό παρακαλώ τον συνάδελφο Σάλμπα να αναζητήσει συμβιβασμό στο θέμα αυτό που θα συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους. Εμείς πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα στην ε, πολιτική μας ομάδα και συμφωνώ και με αυτό που πρότεινε περίπου ο κύριος Γκοσές, ο συντονιστής μας. Κατόπιν τούτου παρακαλώ στις ε, συναντήσεις των ε, σκιωδών ε, εισηγητών να μην προβλεφθούν πάλι εξαιρέσεις. Κάποιοι 6-7 λαμβάνουν αποφάσεις επειδή υποτίθεται έχουν πίεση χρόνου τις υποβάλλουν μόνο στα αγγλικά και μετά μας λένε ψηφίστε. Εγώ νομίζω ο συνάδελφος Κλούτε μας ε, παρουσίασε λιγάκι τις ε, διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριγωνικού διαλόγου με την ελληνική προεδρία όπου η αριστερά πλευρά πρόκειται να δεχτεί κάποιες ύποπτες προτάσεις του Συμβουλίου και εγώ είπα κάθε τράπεζα, μα κάθε τράπεζα για λόγους μη διακριτικής μεταχείρισης να προσφέρει ένα βασικό κανονισμό. Και στην περίπτωση αυτή ο συνάδελφος Κέμπαν είπε εγώ είμαι ο καθαρόαιμος μαρξιστής και όχι ο κύριος Κλούτε και είμαι πάρα πολύ περήφανος που εγώ υπερασπίστηκα πραγματικά τα συμφέροντα του καταναλωτή και όχι των τραπεζών. Okay. Um, I think we've got some interesting repartee, but have you finished, Werner? Yes. Ενδιαφέροντα επιχειρήματα, δεν ξέρω αν τελείωσες. Jean-Paul Gauzes. Jean-Paul. Gauzes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από την παρουσίαση του Βέρνερ Λάγκεν, Βλέπουμε ότι η διάρκεια στο Κοινοβούλιο δεν αφαιρεί ικανότητα δράσης. Θα είμαι σύντομος να πω στους δύο εισηγητές ότι τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ. Πόσο μάλλον που ήμουνα και ο πρώτος εισηγητής στην προηγούμενη εντολή και ξέρω ότι είναι σκληρή αυτή η δουλειά, περίπλοκη, τεχνική και του συγχαίρω για τις προτάσεις τις οποίες μας έκανα. Να υπενθυμίσω αυτά που λέγω από το 2006 για τις πληρωμές. Η πληρωμή είναι μια εμπορική δραστηριότητα, είναι χρήσιμη μεν αλλά εμπορική δραστηριότητα. Σαν τέτοια οι εταιρείε που συμμετέχουν αλεξαρτήτως του καθεστώτος τους πρέπει να αμείβονται δίκαια. Και γι' αυτό και συμφωνώ με τις προτάσεις οι οποίες έγιναν από το ΒΕΝΑ και άλλους έτσι ώστε ε, να γίνει μια οικονομική πραγματικότητα η προμήθεια για τις ε, συναλλαγές με κάρτες, να είναι μια υπηρεσία, σε πραγματι... μια αμοιβή για πραγματικά παρεχόμενη υπηρεσία, ανάλογα βέβαια με το ύψος της συναλλαγής κτλ. Να ακολουθήσουμε λοιπόν τις προτάσεις του εισηγητή για τις ε, προμήθειες αυτές και να μην λέμε ας καταργήσουμε τις, α, τις αμοιβέ τις προμήθειες γιατί αυτό θα είναι φθηνότερο. Δεν θα βοηθηθούν πολύ και δεν θα ωφεληθούν οι καταναλωτές από αυτό. Και αν δεν πληρώνουμε αυτούς που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα θα είναι πιο φθηνά άμα επεκτείνουμε αυτή τη λογική. Πρέπει λοιπόν οι εμπλεκόμενοι στις οικονομικές συναλλαγές να αμείβονται δίκαια για τη συμμετοχή τους. Κατά τα άλλα νομίζω ότι οι συμβιβαστικές προτάσεις είναι ενδιαφέρουσες. Ένα σημείο, μία τροπολογία την οποία υποστήριξε ο Μπεσέ προηγουμένως. Είχα καταθέσει μια τέτοια τροπολογία και την απέσυρα. Γιατί την απέσυρα. Είδα και αναφέρομαι στην τροπολογία για τις μικρές πληρωμές με ε, το τηλέφωνο. Αυτές ε, οι εξαιρέσεις πρέπει να συνεχιστούν γιατί αλλιώς θα παραλύσουμε έναν τύπο δραστηριότητας χρήσιμο για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τις διαδικασίες πληρωμών ε, από τις τράπεζες δεύτερου τύπου. Και γι' αυτό απέσυρα την τροπολογία μου και καλό και τον συνάδελφο Μπεσέ να το ξανασκεφτεί. Ευχαριστώ. Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τα μπλέξαμε λίγο για τους σκιώδεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ εκπροσωπώ την Ιντβελτ τώρα. Τώρα, 0,1 ε, ε, για τις πιστοτικές κατάργηση για τις άλλες, ε, ένα έτος μεταβατική περίοδο για εξίσωση με εσωτερικές συναλλαγές, εξαίρεση των, των προγραμμάτων τρίτου τύπου, co-badging, υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξαιρέσεις κατηγοριών από την εμβέλεια των κανονισμών. Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της σκιώδους εισηγήτριας. Οι σκιώδεις κανονικά ακούγονται στην ομάδα μας, θα δούμε τι θα επικρατήσει στο τέλος. Άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Λάγκεν γιατί μου έδωσε την εντύπωση ότι και σε κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες υπάρχουν προβλήματα, όχι μόνο στη δική μου. Εγώ παλεύω με τη συνείδησή μου του φιλελεύθερου βουλευτή γιατί πάντα ήμουνα κατά του ανωτάτου ορίου. Κάθε τύπου ανετάτου ορίου δεν είναι καθήκον δικό μας αυτό, είναι θέμα αγοράς. Αλλά θα δεχθώ σε αυτές τις συνθήκες ε, μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο καθορισμό ανωτάτου ορίου. Όλοι έχουμε δυσκολίες λοιπόν κύριε Λάγκεν. Για τον φίλο Νίλς σχετικά με τις μικροπληρωμές. Αυτό είναι σοβαρό θέμα και ελπίζω να καταλήξουμε κάπου. Στην ΙΝΚΟ χτες ψηφίσαμε ε, κάτι που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να βάζουν ε, χαμηλότερα εθνικά ανώτατα όρια μέσω των δικών τους αρχών ελέγχου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ε, καλύψουμε τις ανάγκες των συναδέλφων έτσι όπως ακούστηκαν και χτες. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Βέβαια πρέπει να καθορίσουμε ότι οι μικροπληρωμές θα πρέπει να έχουν χαμηλότερο ανώτατο όριο. Ακόμα και χαμηλότερο από τα 12 δολάρια που ισχύει στη ΣΥΠΑ σε κάποιες τουλάχιστον από τις χώρες μας, σε κάποιες από τις χώρες μας απαιτείται να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Μάριαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ως θέμα αρχής είμαι υπέρ μιας ελεύθερης αγοράς με πλήρη ρόλο του ανταγωνισμού. Αλλά εδώ το πρόβλημα που υπάρχει πολλά χρόνια με πείθη για το ότι η Κομισιόν κάνει αυτή την πρόταση για ανώτατο όριο. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο. Έχω καταθέσει και μερικές τροπολογίες που αφορούν <clears throat> πρώτον τις χρεωστικές κάρτες γιατί νομίζω ότι η προμήθεια που πληρώνουμε για αυτές πρέπει να γίνει μηδέν. Έχουμε ήδη εγκρίνει νομοθεσία που χορηγεί τέτοιες χρεωστικές κάρτες για όλους και δεν μπορούμε η Διατραπεζική Επιτροπή να υψώσει όρια. Δεύτερη τροπολογία που έχω καταθέσει, τα όρια ή μάλλον η αποδοχή όλων των καρτών. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα άρνησης των ακριβών καρτών από τους εμπόρους. Γιατί διότι είναι και αυτός ένας παράγων ανταγωνιστικότητας. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει όσο το δυνατόν να παίξει το ρόλο του ο Εκτός αυτού, εκτός αυτού λέγω, τίθεται το εξής θέμα ένας έμπορος μπορεί ή όχι να αρνηθεί κάποια κάρτα. Και εδώ ορισμένοι περιορισμοί να υπάρχει ένα περιθώριο λιγμών του εμπόρου να μπορούν να μην τις δεχτούνται όλες τις κάρτες δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να δεχτούν κάρτες που έχουν πιο ψηλό κόστος για εκείνους από ότι αυτές που χρησιμοποιούν ήδη. Όσο για το co-budgeting, Έχω και εγώ καταθέσει μερικές τροπολογίες κυρία Πρόεδρε για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Σωστά είναι τα προτινόμενα αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες για να είμαστε βέβαιοι ότι ο καταναλωτής ή ο έμπορος θα ξέρει τι ακριβώς ισχύει. Ζητώ λοιπόν από τον εισηγητή να λάβει υπόψη του και τις τροπολογίες αυτές και τον ευχαριστώ για όσα έκανε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν επέστρεψε ο Γουλφ ακόμα. Ο Πάμπλο λέει ότι δεν θέλει πολύ χρόνο για να απαντήσει, άρα ας ακούσουμε την Κομισιόν, όχι πολύ όμως τώρα, όχι πολύ ώρα. Και να ακούσουμε και απαντήσεις λοιπόν. Ορίστε κυρία Κομισιόν μου. Και εγώ σύντομη θα είμαι, αλλά συγχαίρω πράγματι για την ποιότητα των τροπολογιών που δείχνουν μεγάλη γνώση της αγοράς. Uh, uh, και νομίζω ότι έτσι θα καταλήξουμε σε πολύ σωστου συμβιβασμούς. Λοιπόν, ένα θέμα είναι το ύψος των προμηθειών, το άλλο είναι τι συμβαίνει όταν χαθούν οι κάρτες και τρίτον η διαφάνεια κατά τη μεταβατική περίοδο. Τώρα για το κόστος που εφαρμόζουν οι εταιρείε καρτών. Δεν αφορά αυτό τα συγκεκριμένα ποσά γιατί συζητήσαμε ήδη στην αξιολόγησή μας τι αποτελέσματα θα είχε η εφαρμογή των προτινομένων προμηθειών ή εισφορών και θα θέλαμε να μάθουμε και πώς υπολογίζεται το κόστος αυτό, πώς παίζει εδώ ο ανταγωνισμός και όπως γνωρίζουν πολλοί βουλευτές υπάρχει μια μελέτη που ακόμα δεν τελείωσε για το κόστος με το οποίο βαρύνεται ο έμπορος. Και κατά τη διάρκεια της μελέτης λάβαμε πολλά αιτήματα να επιδείξουμε ανοιχτό πνεύμα. Και Συνεχίζεται λοιπόν η μελέτη και θεωρούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε παρά κατά τον Ιούνιο. Υπάρχουν όμως ήδη μερικά προκαταρκτικά συμπεράσματα και ελπίζουμε να κάνουμε μία παρουσιασούλα τους σε μία εκδηλωσούλα την επόμενη εβδομάδα. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε την ανακοίνωση που αφορά αυτή την ε, παρουσίαση στην ιστοσελίδα μας. Θα γίνει και μια παρουσίαση που θα δημοσιευτεί κιόλας. To Και νομίζω ότι θα αναφέρει και τι υπάρχει ως διαφάνεια και τι χρειάζεται ακόμη να εφαρμοστεί. Μετά, αν οι εταιρείε καρτών χάσουν κέρδη από, ως αποτέλεσμα της πρότασης. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Και αυτό φαίνεται από το ότι υπάρχουν χώρες όπου δεν εφαρμόζονται διατραπεζικά κόστη και όμως υπάρχει μεγάλη άνθηση των δοσοληψιών με κάρτες. Τώρα για τις χρεωστικές κάρτες πολλές μελέτες δείχνουν ότι η χορήγηση καρτών αποφέρει μεγάλα κέρδη στις τράπεζες, πολύ ψηλότερα από ό,τι σε άλλους τομείς τραπεζικούς ή της οικονομίας όπως τι λιανικές πωλήσει. Υπάρχει και μια απόφαση του δικαστηρίου όπου το δικαστήριο τόνισε ότι η χρησιμοποίηση καρτών ε, αποφέρει και πρόσθετα κέρδη όπως επιτόκια. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτό να βλάψει τις τράπεζες και φυσικά τα ωφέλη από τη χρήση της κάρτας μπορεί να διαφέρουν από κάρτα σε κάρτα ή από εποχή σε εποχή γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι οι καταναλωτές πάντα όλες τις κάρτες που διαθέτουν. Όσο για τη διαφάνεια έχει υπάρξει συζήτηση για τον διαχωρισμό με το co-badging το μόνο που θα έπρεπε να τονίσουμε ως Κομισιόν είναι ότι εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις προτάσεις, μεταξύ άλλων και γιατί θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Αν χρειαστούν ακόμη τέσσερα χρόνια και φανεί ότι χρειάζεται η περίοδος αυτή, αν καταλήξουμε σε πιο αποτελεσματική αγορά, τότε μπορεί να μην χρειάζεται πια να βάζουμε αυτά τα cap fees. Τέλος για τη μεταβατική περίοδο. Εδώ έκανα μια έρευνα γιατί βέβαια η συζήτηση είναι αν θα πρέπει να είναι μονοετής, διετής. Στο παρελθόν η κάρτα Visa απαιτεί την αποπληρωμή σε δύο μήνες. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις σε δέκα μήνες. Η Mastercard τέσσερις μήνες στη Γαλλία. Μειώνονται τα κόστη και για τις χρεωστικές και για τις πιστοτικές κάρτες μετά από τρεις μήνες και για τη Visa και τη Mastercard δύο μήνες, το είπα και πριν. Τέλος, υπάρχουν τρεις χώρες μέλη που ήδη έχουν νομοθεσία μείωσης των εισφορών στην Πολωνία ας πούμε που εφαρμόζει εξαμηνιαία μεταβατική περίοδο, Πολωνία ναι, και Ρουμανία. Η δεύτερη, η δεύτερη, είπα, η δεύτερη είναι η Ρουμανία. Έξι μήνες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ουγγαρία, αλλά οι δύο χώρες μέλη που ήδη εγκρίνουν αυτή τη μεταβατική περίοδο μείωσης του κόστους είναι αυτές που είπα. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας. Διακόπτει η κυρία Μπάουλς. Κανονικά όταν ζητάς το λόγο μιλάς πολύ. Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα. Ε, πράγματι και οι δύο εισηγητές έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να καταθέσετε τις συμβιβαστικές σας λύσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για να τα συζητήσουμε στις πολιτικές μας ομάδες την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Βέρνερ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα σε καλοδεχτούμε στην επόμενη συνάντηση των εισηγητών που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα λάβουμε υπόψη αυτές τις προτάσεις που έχεις κάνει. Συμφωνώ μαζί σου ότι το 0% για την ανώτατη προμήθεια. Είναι κάτι που δύσκολα θα τύχει η συμβιβαστική πρόταση. Νομίζω λοιπόν ότι σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε πρέπει να υπολογίζουμε στην ε, συμβιβαστική διάθεση όλων των εισηγητών. Κατατέθησαν και συγκεκριμένες προτάσεις, ε, όπως επίσης συγκεντρώσαμε και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας και τους σκιώδεις και τους συζητητές. Να διευκρινίσω κάτι προς τον κύριο Λάγκεν για τις συμβιβαστικές προτάσεις. Δεν είναι τελικές συμβιβαστικές αυτές οι τροπολογίες, είναι προτάσεις συμβιβαστικές. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτές τις προτάσεις και δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα γιατί αυτό θα δημιουργούσε κάποιο χάος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που είναι πάντα ανοιχτές. Σχετικά με το co-badging τώρα, την κοινή το κοινό εταιρικό ή εμπορικό σήμα. Ε, εδώ θα ήθελα να υπάρξει μια κάποια ευελιξία στα πλαίσια του κομπάντζινγκ έτσι ώστε ένας καταναλωτής να μπορεί να προεπιλέξει το σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει για να πληρώσει έτσι ώστε να υπάρχει και ευελιξία και αποτελεσματικότητα στο σύστημα. Σχετικά με τον κανόνα αποδοχής όλων των καρτών. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον έμπορο να επιλέξει εδώ η δυνατότητα αυτή του εμπόρου θα έχει σαν στόχο μόνο τις κάρτες οι οποίες είναι εκτός πλαισίου αν θέλετε προβλεπομένου από την πρόταση και όχι αυτές οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πρότασης στόχος μας είναι να έχουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό, ένα σύστημα ασφαλές, αλλά για τις κάρτες που είναι εκτός είναι απαραίτητο ο έμπορος να έχει μια ανταμοιβή γι' αυτό. Τα υπόλοιπα θέματα θα τα συζητήσουμε πάλι και την επόμενη εβδομάδα, εφόσον δεν έχουν αντίρρηση και οι υπόλοιποι σκιώδεις. Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για την συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για να προχωρήσουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και ιδιαίτερα τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ Παύλο. Ο Ντιόγκο είναι τελευταίος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Σάρων. Εγώ θα ξεκινήσω υπογραμμίζοντας τον θετικό τρόπο με τον οποίο ε, διεξήχθη η συγκεκριμένη συζήτηση και συνεχίζεται η συζήτηση. Για το δύο δεν άκουσα πάρα πολλές ε, πολεμικές ε, αντιπαραθέσεις. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία δεν δημιουργεί πάρα πολύ ενδιαφέρον και όχι και πάρα πολλές αντιδράσεις. Είναι όμως όλες οι οδηγίες γύρω στο συγκεκριμένο κλάδο, από το συγκεκριμένο κλάδο, σημαντικές. Είναι κάτι το οποίο άπτεται φυσικά του ευρύτερου προβληματισμού για τον ανταγωνισμό. Ξέρουμε ότι από τις ρυθμίσεις αυτές θα εξαρτηθεί αν η κατάσταση στην αγορά. Και οι ισχυώδεις εισηγητές αυτό θέλουν να πούν. Ότι εμείς βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και μπορούμε να καταλήξουμε αρκετά γρήγορα σε καλές συμφωνίες. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι μπορεί να πάρουν αύριο στις 8 στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Όσοι μπορεί να είναι παρόντες είναι καλοδεχούμενοι. Ε, όταν καταλήξουμε στις συμβιβαστικές προτάσεις τις τελικές θα τις διανύμουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα ξεκαθαρίζει αρκετά τα πράγματα ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίσαμε. Αυτό το οποίο δημιουργεί πάντα κάποια θέματα είναι οι λεγόμενες υπερτιμολογήσεις. Κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις και κάποια επιπλέον οικονομικά βάρη. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να δημιουργήσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού αν υπάρχει μια συναλλαγή ε, τετραμερής, βέβαια τα πράγματα περιπλέκονται σε σχέση με την τριμερή συναλλαγή. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε και εγώ και οι συνεισηγητές να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Και το είπαν και αρκετοί από τους προλαλήσαντες, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Συμφωνία η οποία να είναι κατανοητή, απλή, δεν υπάρχει μία άποψη και μία θέση σε σχέση και με το θέμα των υπερτιμολογήσεων. Οι προτάσει τι οποίε μα έχει καταθέσει το συγκεκριμένο τομέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζουν και κάποιε αδυναμίε εφαρμοστικά. Το θέμα αυτό έχει σαν στόχο το να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στους εμπόρους στα πλαίσια των τριμερών συναλλαγών. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση η οποία να είναι εφαρμόσιμη στο σύνολο των ειδικών καταστάσεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι έχω πράγματι εμπιστοσύνη στο ότι θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε στις 20 Φεβρουαρίου και αυτές τις τροπολογίες και την υπόλοιπη έκθεση. Νομίζω επίσης ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην Ολομέλεια το μήνα Απρίλιο Ό,τι ακούω από τους συναδέλφους σκιώδης προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται. Επ' αυτού λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τερματίσει την εντολή του την παρούσα περίοδο με την αίσθηση ότι κάτι πέτυχε. Γι' αυτό και άλλωστε έχουμε εκλεγεί. Σας ευχαριστώ όλους. Πρόκειται. Θα ψηφίσουμε στην οίκονη τότε που σας είπα για να φτάσουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου 1. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο, στα σημεία 6, 7 και 8 τις απαλλαγές δηλαδή του 12 όσοι φεύγουν παρακαλώ να φεύγουν ηρέμως διότι αλλιώς δημιουργείται σύγχυση. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Γι' αυτό παρακαλώ να φεύγετε, αποσύρεστε ηρέμως. Αντουλίν, είσαι έτοιμος? Σε muchas gracias. Comienzo. Sí. Muchas gracias, presidente. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε εξετάζουμε τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατοθεί στις ε, γνωμοδοτήσεις για τις απαλλαγές των τριών αρχών. 34 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Οι 34 αυτές για μια στιγμή λέει η πρόεδρος διακόπτη τον κύριο Σάντσες Πεσέδο. Παρακαλώ να μην συζητάτε, έχουμε ξεκινήσει ε, άλλη συζήτηση τώρα ιδιαίτερα πίσω από τον εισηγητή, στις πλάτες του εισηγητή. Συνεχίζει ο κύριος Πεσέδο λοιπόν. Έχουν κατατεθεί 34 τροπολογίες και για τις τρεις αρχές. Για μία 11 και για τις άλλες λιγότερες. Οι ίδιοι έχουν καταθέσει τις τροπολογίες σε όλες τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού και για τα τρία όργανα. Τις περισσότερες από τις τροπολογίες τις δέχομαι γενικά. Δέχομαι επίσης τις εργασίες τις οποίες έχει, ε, έχουν προτείνει οι συνάδελφοι. Ίσως θα ήθελα να ακούσω και από πλευράς αυτών που καταθέτουν τις τροπολογίες για να τις σχολιάσω μετά. Αλλά πάντως όπως σας είπα, γενικότερα οι τροπολογίες αυτές ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές. Κάποιες άλλες ίσως λιγότερα. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τις απόψεις αυτών που καταθέτουν τις τροπολογίες και να τις σχολιάσω ίσως μετά. Ευχαριστώ Αντολίν. Σε αυτή την περίπτωση περνάω στους Σκιώδης. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος ε, και η σημασία, πόσο μεγάλη είναι η σημασία αυτών των απαλλαγών. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε το περιεχόμενο αυτών των απαλλαγών. Εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες και για τις τρεις. Καταρχήν πιστεύω ότι οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν ένα θαυμάσιο σημείο εκκίνησης και παράλληλα θεωρώ ότι πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο ότι οι εποπτικές αρχές ε, βρίσκονται ακόμα εν τη γενέση τους. Άρα δηλαδή αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει καλύτερο συντανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι άλλο που αφορά τις ε, τροπολογίες μου. Εγώ αναφέρομαι στις ε, προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για να υπάρξουν διορθώσεις και θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες ε, ελλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία των εποπτικών αρχών. Παραδείγματο χάρη η εξωτερική ανάθεση των ε, συστημάτων πληροφορικής τα θέματα των δημόσιων διαγωνισμών και επίσης και οι διαδικασίες ε, επιλογής, η διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής. Έχω συμπεριλάβει και ένα νέο στοιχείο το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού. Ε, το πώς αυτό πρέπει να προβλέπεται ε, στους προϋπολογισμούς. Αυτό αφορά και τις τρεις εκθέσεις. Επίσης, θεωρώ ότι επειδή αυτές ε, οι αρχές βρίσκονται, όπως σας είπα, εν τη γενέση τους, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αποκτήσουν περισσότερες αρμοδιότητες και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τους προσφέρουμε και περισσότερους πόρους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ίσως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να αναζητήσουμε ε, κάποια αναδιοργάνωση ή κάποιες ε, άλλες δυνατότητες ε, για να είναι πιο αποτελεσματικές. Και αν συμβεί αυτό, τότε προφανώς θα πρέπει να υπάρξει κάποια αύξηση στους προϋπολογισμούς. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, πρέπει να σας πω ότι είδα τις τροπολογίες και διαπίστωσα ότι Κάποιοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει περίπου τις ίδιες ε, τροπολογίες με μένα και συμφωνώ ότι το μεικτό σύστημα χρηματοδότησης ε, ε, δεν είναι το καλύτερο. Πρέπει να αναδιαρθρωθεί είτε να προβλέπεται μια ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό ή κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει χρηματοδότηση από εισφορές που θα επιβληθούν στην αγορά. Και βεβαίω, μέσω των συμβαστικών προτάσεων μπορούμε να διευκρινίσουμε λιγάκι τι ακριβώς εννοούμε. Σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με τις ε, τροπολογίες που έχουν ε, καταθέσει οι συνάδελφοί μου όσον αφορά τους προϋπολογισμούς. Λίγες είναι σχετικά οι τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι ε, ακολουθούν όλες την ίδια κατεύθυνση και κατόπιν τούτου δεν θα είναι δύσκολο να αναζητήσουμε συμβιβασμούς. Και όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει για τους ε, συμβασμούς, με μεγάλη μου χαρά να βοηθήσω τον εισηγητή στη δουλειά του. Πρόεδρος Ιάν Γένσεν, εκ μέρους των Φιλευθέρων δεν μπορεί να παρίσταται. Ε, Μου έστειλε βέβαια ένα σημείωμα ε, που λέει ότι καταθέτει κάποιες τροπολογίες, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνεί με την εισηγήτρια. Δεν ξέρω, μήπως σας έχει δώσει εσάς κάποιο σημείωμα. Όχι, αλλά έχουμε υπογράψει τις ίδιες ε, τροπολογίες και οι τρεις μας και οι τροπολογίες μας αφορούν τη γραμμή στον προπολογισμό για όσους συμμετέχουν στην αγορά. Ο Σπεν δεν είναι εδώ, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Άρα δηλαδή η γραμμή του προϋπολογισμού φαίνεται να είναι κάτι που σας απασχολεί, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, αλλά θα έλεγα ότι το πιο ακαθόδες θέμα είναι ακριβώς αυτό που δημιούργησε τις περισσότερες ε, τροπολογίες από τέσσερις ομάδες. Τρεις στις τέσσερις τροπολογίες αυτό το θέμα ανέφεραν. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε και εμείς. Γι' αυτό και εγώ το αναφέρω πρώτο. Δεν νομίζω ότι οι τροπολογίες που προτάθηκαν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Μπορούμε να τις συνδυάσουμε και να έχουμε συμβιβασμούς. Μπορούμε. Ξέρουμε βέβαια ότι τα κράτη-μέλη έχουν εισφορές στον προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης δηλαδή Αναρωτιέμαι αν είναι καλή ιδέα αυτή και αν δεν θα έπρεπε στο μέλλον να κινηθούμε προς καθαρά τον ενωσιακό προϋπολογισμό ανεξάρτητα από τα κράτη τώρα. Άλλο θέμα είναι να προέρχονται όλα από τον προϋπολογισμό ή και ένα τμήμα από την αγορά. τρίτη πτυχή του θέματος που δεν έχει αναφερθεί. Για δύο από τα όργανα δεν είναι θέμα, αλλά για το τρίτο είναι. Και πρέπει να δούμε τη δυνατότητα διαφορετικών θέσεων ή γραμμών του προϋπολογισμού. Πάντως η θέση μας ανέκαθεν αυτή ήταν μετά τις νέες δυνατότητες που μας δίνει η απόφαση για το ΕΑΚΑ του δικαστηρίου. Ildiko Ο η Ildiko Γκαλπάλτς είναι η σκιώδηση αρμόδια και αναφέρθηκε στην αύξηση της χρηματοδότησης μια αύξηση της χρηματοδότησης η οποία θα επιτρέψει να προχωρήσουν οι εργασίες αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχει μηχανική αύξηση αλλά να υπάρχει ανταπόκριση με τις πραγματικές ανάγκες. De autoridad en fase de implantación y establecimiento. Μιλάμε για μια δυνατότητα που πρέπει να δώσουμε εμείς για διευκόλυνση της εγκατάστασης αυτής της αρχής όπως επίσης και σωστού καθορισμού των νέων αρχών, και, των αρχών αυτών και των νέων ευθυνών τις οποίες αναλαμβάνουν. Αυτή πρέπει να είναι η βασική γραμμή. Οι αυξήσει να μην είναι μηχανιστικές αλλά να ακολουθούν μια λογική εφόσον είναι πράγματι απαραίτητες. Αυτή είναι η βασική γραμμή και θα προσπαθήσω να καταθέσω μια συμβιβαστική λύση, πρόταση γι' αυτό. Υπάρχουν και ορισμένες τροπολογίες οι οποίες είναι λογικές και μπορώ να τις δεχτώ. Αυτές οι οποίες ε, έχουν σχέση τις διορθώσεις για το ελεγκτικό συνέδριο. Θέματα όπως οι δημόσιοι διαγωνισμοί, το outsourcing, ε, και μια μεγαλύτερη διαφάνεια γενικά στον τρόπο λειτουργίας και στον υπολογισμό του κόστους αυτού του τρόπου. Και εδώ εγώ υποστηρίζω τις τροπολογίες αυτές, δεν χρειάζονται εδώ να υπάρξουν συμβιβαστικές, χρειάζεται μια απλή θετική απόκριση. Ο κύριος Μάρτιν κατέθεσε και αυτός τροπολογίες, δύο από αυτές αναπαράγουν ουσιαστικά κάποια θέματα τα οποία <clears throat> αναφέρονται σε προηγούμενες απαλλαγές όπως επίσης και το θέμα του κόστους των ενοικίων θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία γύρω από τα θέματα αυτά και επίσης το θέμα του, ε, των δικτών κόστους για τις μεταφράσεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο όχι σε επίπεδο διατύπωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει μου δημιουργεί ένα με κάποιο πρόβλημα, γιατί νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι αυτό το οποίο λέει ότι από πλευράς των αρχών θα ζητήσουμε να αποφευθεί η γραφειοκρατία και η επιβάρυνση γενικά. Το θέμα είναι ότι αυτές οι αρχές ε, οι οποίες λειτουργούν φυσικά σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών όταν θέλουν να συλλέγουν πληροφορίες προφανώς στρέφονται στις ομόλογες αρχές τους σε εθνικό επίπεδο. Η εποπτεία ακριβώς συνίσταται στο να συλλέγουν πληροφορίες και αυτό δεν είναι ένα επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος, είναι βασική λειτουργία των δημοσίων αρχών και των εποπτικών αρχών, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και η δραστηριότητα αυτή και σε οικονομικό επίπεδο θα είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμη. Αλλά αυτή η τροπολογία νομίζω ότι μου δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες γιατί στην ουσία αντιτίθεται στο να συλλέγουν τις πληροφορίες τις οποίες επιθυμούν και χρειάζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Κατά τα άλλα πάντως αντιμετωπίζω θετικά τα υπόλοιπα θέματα. Σημερίζομαι λοιπόν με τις υπόλοιπες τροπολογίες. Πρόκειται για μια προσπάθεια συνολική. Εκπροσωπούνται όλες οι ευαισθησίες και όλες οι απόψεις. Δεν εισάγονται στοιχεία μέσω των τροπολογιών αυτών που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομική επάρκεια και την λειτουργία των συγκεκριμένων αυτών και για, ε, υπηρεσιών και πρέπει να γίνουν δεκτές. Ίσως θα υπάρξουν κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις γιατί πάνω στα ίδια θέματα θα αντιμετωπίζονται από τις πολιτικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο και θα προσέξουμε έτσι ώστε η τελική πρόταση να είναι όσο πιο εναρμονισμένη γίνεται. Ευχαριστώ. Στοχεύουμε λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε στις 20 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Ελέγχου και να φτάσουμε στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Το επόμενο θέμα αφορά την Τρόικα. Δεν βλέπω τους εισηγητές. Θα έπρεπε να είχαν έρθει αλλά θα διακόψουμε για πέντε λεπτά. Να έρθουν οι εισηγητές για την Τρόικα, για το θέμα της Τροίκης. Ναι. Madame Pérez. Thank you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

Okay. Um, right, we're, we're, we're, we're here now. Um, λοιπόν, τώρα περνάμε στη δική μας έκθεση περί της Τροίκης για την Τρόικα με τον Ότμαρ Καράς και τον κύριο Νγκόκ. Ε, υποβλήθηκαν πολλές τροπολογίες, μερικές τις κατέθεσα και η ίδια. Θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές πρώτα και μετά ο συνήθως θα περάσουμε στους σκιώδεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο Ότμαρ πρώτος. πρώτος. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Συνησυγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε γιατί έχουν κατατεθεί τόσες πολλές τροπολογίες. Κατά τη δική μου άποψη αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι καταθέσαμε σχέδιο έκθεσης για να δρομολογηθεί η διαδικασία πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας και πριν ξεκινήσουν και οι ακροάσεις. Το κάναμε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα ερωτηματολόγια και με βάση τις απαντήσεις θελήσαμε να έχουμε τη βάση της δουλειάς μας. Έκτοτε βέβαια έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι. Έχουμε κάνει νομίζω περίπου έξι ακροάσεις. Έχουμε κάνει τέσσερα ταξίδια και εντωμεταξύ έχουμε αξιολογήσει και τα ερωτηματολόγια και νομίζω ότι όλοι μας πλέον ε, είμαστε πολύ καλύτερα ενημερωμένοι, έχουμε μια πολύ πιο ισόρροπη εικόνα, βέβαια ο καθένας μας με τη δική του προσωπική τοποθέτηση. Το σχέδιο της έκθεσης κατατέθηκε στις 17 Δεκεμβρίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι Έκτοτε συμμετείχαν ενεργά στις διάφορες εργασίες που έλαβαν χώρα. Έχουμε 297 τροπολογίες από το ΕΛΚ, 200 από τους σοσιαλδημοκράτες, 86 από τους φιλελεύθερους, 193 από τους πράσινους, 12 από το κόμμα των προοδευτικών και της δημοκρατίας, εξίσου επίσης αρκετές από την ΚΟΕ και από τους μη εντεταγμένους. Ε, θα ήθελα να πω κάτι που το είπε ο Λαμπέρ στις ε, αρχές του έτους. Δηλαδή ότι είπε κάτι που και εγώ συμφωνώ 100% ε, με αυτό που είπε. Δηλαδή είπε ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε ευρεία συνένεση με, για αυτή την έκθεση και μόνο η ευρεία συνένεση θα μπορέσει να καταστήσει εφικτές ή εφικτά τα συμπεράσματά μας, τότε λοιπόν σε αυτή την έκθεση επειδή σε 99 ημέρες έχουμε ευρωεκλογές, επειδή υπάρχει αυτό, θα πρέπει να δούμε την πραγματική κατάσταση, να δούμε τα γεγονότα, αυτά να προβάλλουμε. Γεγονότα λοιπόν και όχι ιδεολογική αντιπαράθεση και όχι ιδεολογική ερμηνεία των γεγονότων και των αριθμών. Και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, γιατί στη τελική ανάλυση αυτή ήταν και η εντολή που μας δόθηκε. Στις 12 ε, Δεκεμβρίου αποφασίστηκε στα πλαίσια του χάρτη πορείας να δοθεί μια εντολή για την Τρόικα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, στο πλαίσιο των θεσμών, για τη σχέση των θεσμών μεταξύ τους, για τη δημοκρατική νομιμότητα για τη θεωρητική βάση για τη λήψη αποφάσεων, στατιστικές προβλέψεις, ε, προ, στατιστικές, στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις και ε, κλείνω σε αυτήν την παράθεση που ήταν στα αγγλικά θέλω να πω ότι πάνω απ' όλα αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να εξάγουμε συμπεράσματα αλλά αυτά τα συμπεράσματα θα έπρεπε να βασίζονται στο ενωσιακό δίκαιο και των ενωσιακών μεθόδων. Οι αποφάσεις λοιπόν να λαμβάνονται με βάση αυτά τα δύο στοιχεία γιατί μόνο με το ενωσιακό δίκαιο και μόνο με τις ενωσιακές διαδικασίες μπορούμε να διασφαλίσουμε την διαφάνεια, την ομοποίηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή του χάρτη οικουμενικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων που ο χάρτης αυτός είναι εγγενές στοιχείο των προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, διεξάγονται συζητήσεις ε, ανάμεσα στους ε, συνεργάτες μας, γίνονται συζητήσεις με τους σκιώδης και ελπίζω σύντομα να υπάρξει και άλλη μια συζήτηση ανάμεσα στους συνεισηγητές έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε τη δομή και την ε, μελλοντική διαδικασία. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ομάδες τροπολογιών. Η μία ομάδα αφορά την ανάλυση του γεγονότος ύπαρξης της Τρόικας στα κράτη-μέλη ως ένα τρόπο απάντησης στην κρίση. Αυτή είναι η μία ομάδα. Η άλλη ομάδα αφορά τροπολογίες σε σχέση με τα ίδια τα προγράμματα και νομίζω ότι οι επιπτώσεις των πραγμάτων δεν μπορούν αυτή τη στιγμή ακόμα να αξιολογηθούν ε, σωστά για τα προγράμματα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και τα προγράμματα που σας είπα δεν αποτελούν απαραίτητα τμήμα της εντολής μας. Εμείς βασιζόμαστε στα γεγονότα και θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στοιχεία πριν από την κρίση και τα στοιχεία μετά την κρίση τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να είναι καταλυτικά για τις επιπτώσεις των μέτρων, γιατί εντωμεταξύ μεσολάβησε η μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα σύγκριση στοιχείων. Και οι επιπτώσεις των προγραμμάτων δεν έχουν γίνει ακόμα απόλυτα ορατές. Και θα πρέπει να διερωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν δεν λαμβάναμε κανένα μέτρο, αλλά και αυτό ενδεχομένως να αφορά μελλοντικές εκθέσεις. Εμείς συζητήσαμε διαμακρών σχετικά με τις συνέπειες που προκύπτουν από τις εκθέσεις και αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι ότι πρέπει να οριστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο αφορούν τις περισσότερες τροπολογίες. Και καταλήγουμε στο ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εργαλείο που δεν θα είναι ούτε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, αλλά ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα τροφοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης, γιατί το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είναι νομικά δεσμευμένο να βοηθάει τα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη είναι μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όχι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, για μένα, όσον αφορά στο κέριο ερώτημα που είναι η Τρόικα ή αν θέλετε τα προγράμματα ε, οικονομικής ε, συνδρομής, αυτά πρέπει να τα εντάξουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Βεβαίως ε, και τα, τα κόμματα διαφοροποιούνται ως προς την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Υπάρχει διαφορετική αξιολόγηση και όσον αφορά και την εντολή θα πρέπει να εξετάσουμε την εντολή ως την βάση των συμβαστικών τροπολογιών και υπάρχει και συμφωνία, συνένεση στο ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Διαφάνεια στις ενωσιακές διαδικασίες. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες στις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και οδησηγητές, ποιες μπορεί να είναι οι δομές που θα διέπουν τις συμβαστικές προτάσεις, να εντατικοποιήσουμε τις συζητήσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συμβαστικές προτάσεις που θα καλύπτουν όλα τα κόμματα, όλες τις πολιτικές ομάδες. Ο δικός μας στόχος ήταν και παραμένει να μην κάνουμε μία συζήτηση με αριστερή ή με δεξιά χρειά, αλλά μία συζήτηση που βασίζεται σε γεγονότα, αδιαμφισβήτα γεγονότα. Δεν ε, ιδεολογικοποιούμε τη συζήτηση, αλλά όπως σας είπα βασιζόμαστε σε απλούς ε, αριθμούς, σε γεγονότα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο συνεισηγητής κ. Γκόκ. Ευχαριστώ Σάρων. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου και όλους τους σκιώδεις για όλα όσα κάνανε κατά τις επισκέψεις στα κράτη-μέλη και κατά τις ακροάσεις που κάναμε εκεί όλοι συνεισέφεραν εκεί την αξιολόγηση αυτή του έργου της Τρόικας. Επίσης ευχαριστώ τη γραμματεία που μας, ε, μας ακολούθησε σε αυτόν τον πραγματικό περίπλου την Οδύσσια όπου μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και οι ακροάσεις που κάναμε ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Μια, ένα πρώτο μας καθήκον από κοινού με τον συνεισηγητή ήταν η έκθεση πρωτοβουλίας ή έρευνας, δηλαδή κάτι ενδιάμεσο μεταξύ της Ερευνητικής Επιτροπής και της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτό δικαιολόγησε τους δύο εισηγητές. Και το σχέδιο που παρουσιάσαμε στις 16 Ιανουαρίου ήταν μια ωραία βάση συζήτησης και γι' αυτό ευχαριστώ τον Οτμάρ που προσπάθησε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να γίνει κείμενο αναφοράς κατά τα τέσσερα ταξίδια επισκέψεις που οργανώσαμε. Ενδιαφέρθηκε πολλοί κόσμος. Είναι ισορροπημένο κείμενο και ανταποκρίνεται, αντικατοπτρίζει τις δύο θέσεις κατ' εμέ. Τις θέσεις των δύο ομάδων μας δηλαδή. Ξέρουμε ότι έχουμε διαφορές. Η δική μου ομάδα είχε μια θέση ιδιαίτερα ριζοσπαστική, ιδιαίτερα ο πρόεδρος. Στο ΕΛΚ ξέρω ότι έχετε διάφορες θέσεις, τουλάχιστον τρεις και η δική σας ήταν πολύ απομακρυσμένη από διάφορα συμπεράσματα της πρώτης μορφής του κειμένου με τα οποία συγκλίναμε περισσότερο στη συνέχεια και κατορθώσαμε να κάνουμε εξαιρετική εξισορρόπηση. Το κείμενο δεν είναι καθόλου ιδεολογικό, όπως το είπατε και εσείς ο Αυτός ήταν ο σκοπός, να μην κάνουμε ιδεολογική δουλειά, αλλά αξιολόγηση. Και γι' αυτό θέσαμε τα σωστά ερωτήματα για τους πολλαπλασιαστές, ας πούμε. Τονίσαμε ιδιαίτερα τα ίδια τα επιχειρήματα της Τρόικας και στα τρία της συνθετικά στοιχεία. Εξετάσαμε τους μακροοικονομικούς στόχους που έθεσε και συνεχώς άλλαζε η ίδια η Τρόικα και μετά εξετάσαμε ορισμένες θεσμικές οδούς αρκετά καινοτόμες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε για να δούμε τι θα λέγαμε στις συνεντεύξεις τύπου μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία και ελπίζω η δουλειά αυτή που μας ένωσε τους δύο συνεισηγητές που ως εκπροσώπους των δύο μα ομάδων να παραμείνει η βάση για την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Τι λείπει για να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει η πιο μεγάλη δυνατή πλειοψηφία de Και για την αξιολόγηση της Τρόικας. Γι' αυτό πρέπει εκτός από το σχέδιο που είχαμε υποβάλει να συμπεριλάβουμε και τις θέσεις των σκιωδών. Αυτό μας λείπει ακόμα. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις θέσεις της ΓΚΟΕ, των Πρασίνων, των Φιλελεύθερων και των άλλων ομάδων. Βέβαια, δεν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κείμενο τελείως ε, μπερδεμένο. Πρέπει φυσικά να υπάρχει κάποια συνοχή του κειμένου, αλλά οι τροπολογίες που κατέθεσαν όλες οι ομάδες θα συμπεριληφθούν, θα ληφθούν υπόψη. Μέχρι στιγμής πετύχαμε συμβιβασμό επί 22 παραγράφων μένουν, μένουν λέγω, άλλες 23 τουλάχιστον χωρίς να αναφέρουμε και τις 915 τροπολογίες συνολικά μέχρι στιγμής. Αυτό εξηγεί γιατί εργαζόμαστε τόσο πολύ, γιατί χρειαζόμαστε τόσο πολύ δουλειά, πόσο μάλλον που μάθαμε πολλά εγώ παρατήρησα με τεκπλήξεως κατά τα ταξίδια μας ότι οι τρεις οργανισμοί που αποτελούν την Τρόικα σπανίως έχουν συμφωνήσει. Και γι' αυτό βεβαιώθηκα θέτοντας ερωτήματα σε εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι διαφέρει σε πολλές θέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους για το bail-in ή το bail-out της Ιρλανδίας για τον ρυθμό δημοσιονομικής εξυγένσης κλπ. κλπ. Αυτό εξηγεί γιατί θελήσαμε σε αυτή την τόσο σοβαρή δουλειά να πάρουμε υπόψη μας τα σοβαρά και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν γιατί οι τέσσερις χώρες που εξετάσαμε απαιτούν, δικαιολογούν μια πολύ σοβαρή ανάλυση γιατί οι διαφωνίες μεταξύ των οργάνων της Τρόικας είναι πρόβλημα. Όπως είπατε και εσείς υπάρχει καταρχήν ένα νομικό πρόβλημα της ίδιας της ύπαρξης της Τρόικας, αλλά δεν έχουν συζητηθεί ποτέ και πουθενά στην Ένωση οι διαφωνίες αυτές. Άρα εγκρίθηκαν σχεδόν με το ζόρι, επιβλήθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα democratic accountability στην Ευρώπη που πρέπει να το δούμε δημοκρατικής λογοδοσίας δηλαδή και και πρέπει να το δούμε και αυτό. Τελειώνω θέτοντας ένα ερώτημα προς τον σκιώδη προς τους σκιώδης που θα μιλήσουν σε λίγο έχουμε πολύ στενό χρονοδιάγραμμα αν σκεφτούμε όλα όσα πρέπει να αναλύσουμε για να καταλήξουμε στο πιο στεναρό δυνατό κείμενο για να ακουστούν οι θέσεις μας καθαρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατ' εσάς λοιπόν σκιώδης, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει στην Επιτροπή στις 24 ψηφοφορία αρκεί, σας αρκεί, σας φτάνει. Γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμβιβασμούς μέχρι τότε για να μην τα χαλάσει όλα η ιδεολογική συζήτηση αφού έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε μεγάλη πλειοψηφία για την συμβολική αυτή σημασία έκθεση στο τέλος της θητείας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τους φιλελεύθερους ο Νίλς. Ευχαριστώ να μην έχετε αμφιβολία αυτή τη φορά. Είμαι ο πραγματικός σκιώδης, δεν αντικαθιστώ κανέναν. Λοιπόν, καταρχήν, ευχαριστώ τον Ότμαρ και τον Λιέμ και τους άλλου τους σκιώδης δηλαδή, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Από την πρώτη μέρα με ενδιέφερε και άρα το ερώτημα του στο ερώτημα του Λίαμ απαντάω ναι, ακόμη και αν είναι στενό το χρονοδιάγραμμα, το ενδιαφέρον του θέματος το καθιστά αξίζει τον κόπο να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό ακόμη και αν πιεστούμε. Από πιο θεωρητική άποψη έχουμε τέσσερις πολύ διαφορετικές χώρες τον Κελτικό Τίγρη και την Κύπρο, πολύ ειδικέ περιπτώσεις, πιο ενδιαφέρουσες οι περιπτώσεις της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Νομίζω ότι πληγήκαμε, χτυπηθήκαμε από τρία διαφορετικά κύματα ή προβλήματα. Πρώτον, η παγκοσμιοποίηση ως γενικότερη διαδικασία από το 80-90, ιδίω από το 2000, που έθεσε μερικά προβλήματα. Μετά η δημοσιονομική χρηματοπιστωτική κρίση, που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο στις χώρες αυτές για πρόσβαση στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και μετά το ευρώ. Η περίπτωση του ευρώ είναι πολύ συγκεκριμένη. Αναδρομικά βλέποντας τι αποφασίστηκε ήδη από το 1978 βλέπουμε ότι η σκληρότητα του ευρώ, η ακαμψία του ευρώ είναι, ήταν πρόβλημα από την αρχή της σύλληψής του. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να το δημιουργήσουμε, στην ουσία αποφασίσαμε ένα άκαπτο σύστημα. Κατά τις συζητήσεις της έκθεσης, θέλουμε πάντα να βρίσκουμε τον ένοχο, κάποιον ένοχο. Και σε αυτή την πολύ πολιτική και ιδεολογική συζήτηση είναι δύσκολο να βρεθεί ο ένοχος και γίνεται μερικές φορές η προσπάθεια να αποφύγουμε την ανάληψη εθνικών ευθυνών, η απόδοση εθνικών ευθυνών και σε μια συνέντευξη που έδωσα σήμερα στη Φιλανδία άκουσα ότι η κρίση είναι τεχνητή και οφείλεται στον Όλυ Ρεν. Αυτό είναι όμως δικαιολογία, δεν είναι σωστό. Εύκολο είναι βέβαια να κρύβονται οι πολιτικές ευθύνες βρίσκοντας έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Δεν νομίζω ότι ότι οι τροπολογίες πρέπει να γράφονται με βάση προεκλογικά κριτήρια. Αλλά όμως μερικές από αυτές που έχουν κατατεθεί είναι καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι να καταλάβουμε σε τι βαθμό η Ένωση υπήρξε υπερβολικά αισιόδοξη και δεν είχε λάβει υπόψη της δεόντος τα προβλήματα που υπήρχαν μετά τη Μαύρη Δευτέρα του 97 ας πούμε. Του 87 είπε ο μιλήτης. Κατά τη συζήτηση περί Τρόικας ε, ακούστηκαν και μερικές παραπληροφορήσεις. Η Κομισιόν είχε νομική βάση και νομιμότητα για τη δράση της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και διάφορα προβλήματα που θα έπρεπε να αποφευχθούν στην επόμενη κρίση ή στην επόμενη φάση της κρίσης. Επίσης πρέπει να ξέρουμε τι αποφάσεις πήραμε για το δίμετρο και το εξάμετρο για να αποφύγουμε παρόμοιες κρίσεις. Πολλοί θα πούν ότι αυτά τα μέτρα ήρθαν πολύ αργά. τονίσαμε ότι οι τράπεζες ήταν προβληματικές αλλά δεν είδαμε αν ήταν πρόβλημα και οι διάφορες πολιτικές κοινωνικής περίθαλψης στις διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα ιδίως το σύστημα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πίεση της κρίσης και Γι' αυτό υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωπους εκτός προγραμμάτων υγειονομικής καν περίθαλψης. Η απασχόληση βέβαια αναφέρεται πολλές φορές στις τροπολογίες αλλά Προ στιγμή να στα αφήσουμε για την Επιτροπή Απασχόλησης και την έκθεσή της. Αν στην επόμενη κρίση συνεχίσει η Ευρωζώνη και το Eurogroup να υπάρχει, τότε χρειάζονται ορισμένες αλλαγές είναι υπόλογο στο, προς το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα έπρεπε να είναι ο υπεύθυνος για τη λήψη της τελικής απόφασης. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με το 17 της συνθήκης θα έπρεπε να είναι ο αρμόδιος θεματοφύλακας και η ΕΚΤ να παίζει ρόλο παρατηρητή το δονουτού εάν χρειαστεί να είναι περιθωριακός δανειοδότης συμπληρωματικός. Και τέλος, κάτι για τα διαρθρωτικά ταμεία. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη έλλειψή μας είναι η, πολλα... η πλημελής λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων από πολλά χρόνια ήδη πριν που δεν κατάφεραν να πετύχουν τη σύγκληση που ελπίζαμε. Βλέπουμε οικονομική σύγκληση από το 50, 60 και 70 βλέπαμε και όλοι νόμιζαν ότι θα υπήρχε ένας παράδεισος ευημερία, αλλά από τα μέσα ήδη του 70 είδαμε ότι οικονομικά ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και ότι θα έπρεπε ρίζικα να αλλάξει η λειτουργία των διαφορετικών ταμείων. Έπρεπε να το είχαμε δει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους των Πραστίνων ο Φιλίπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την πολύ καλή τους δουλειά. Εγώ δεν μπόρεσα να συμμετέχω σχεδόν σε καμία ε, επίσκεψη εκτός από την Ελλάδα και εκεί πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Ε, διαβάζει κανείς διάφορα πράγματα, αλλά το να τα δει κανείς και επιτόπου είναι διαφορετικό. Όσον αφορά την την έκθεση, όπως είπε και ο Ότμαρ, εγώ τάσαμε υπέρ μιας έκθεσης που θα εγκριθεί με όσο δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία. Αλλά όχι όμως με το τίμημα του τελικά να μην τίποτα. Ξέρω βέβαια ότι αυτό δεν είναι το στυλ του εισηγητή. Ξέρω ότι είμαστε σε καλά χέρια και πρέπει λοιπόν η έκθεση να είναι όσο πιο συγκεκριμένη και προχωρημένη γίνεται. Ξέρω ότι υπάρχει ο πειρασμός ε, να συζητήσουμε για τη δημοκρατική λογοδοσία, κυρίως για το θεσμικό στοιχείο της λογοδοσίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε το όλο θέμα, γιατί πιστεύω ότι εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και θεσμοί οι οποίοι τάσσονται υπό την αιγίδα του ενωσιακού δικαίου, εφόσον συμβούν αυτά, τότε έχουμε περισσότερες δυνατότητες να εφαρμόσουμε πολιτικές, οι οποίες ε, θα γίνονται περισσότερο θα σέβονται περισσότερο το χάρτη των ε, ανθρωπίων δικαιωμάτων και θα οδηγούν σε καλύτερη ισορροπία. Έτσι λοιπόν ξέρω ότι και το θεσμικό στοιχείο επηρεάζει πάρα πολύ τις ε, πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Αυτών όλων λεχθέντων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πολύ τίμια και ειλικρινά αυτά τα οποία συνέβησαν. Ελέγχθησαν πάρα πολλά για το μακροοικονομικό στοιχείο της κρίσης. Νομίζω όμως ότι θα ήταν λάθος αν αυτή η Επιτροπή αγνοούσε ή αν άφηνε απλά την Επιτροπή Επασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να ασχοληθεί αυτή μόνο με το θέμα των ανισοτήτων, την στέρηση κοινωνικών δικαιωμάτων και αυτό για δύο λόγους το πιστεύω. Δεν θέλω αυτή η Επιτροπή να εκλαμβάνεται ως ε, η Επιτροπή των Αριθμών, των μανιακών με αριθμών που απλά ενδιαφέρονται για μακροοικονομικά αποτελέσματα και ξεχνάνε ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Εγώ δεν πιστεύω ότι με τους ανθρώπους ασχολείται η Επιτροπή Απασχόλησης και με τους αριθμούς η Επιτροπή δική μας. Κάθε άλλο. Εμείς εξετάζουμε το οικονομικό θέμα και τι υπάρχει πίσω από την οικονομία. Γιατί τελικά η οικονομία υπηρετεί τους ανθρώπους. Αυτό είναι καθαρά πολιτικό, πολιτική ερμηνεία το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει σε πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε μεγαλύτερη ανισορροπία ή σε λιγότερη ε, υγειονομική κάλυψη ή σε μικρότερη κοινωνική κάλυψη, τότε η σε λιγοτερη υγειονομικη καλυψη η δυνατότητα της οικονομίας να προσφέρει ευημερία μειώνεται. Άρα δηλαδή μιλάμε για άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Κατά τη δική μας άποψη, μια κοινωνία που είναι ε, σε καλή κατάσταση δεν είναι το αποτέλεσμα μιας εύρυθμα λειτουργούς οικονομίας, αλλά είναι η προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά η οικονομία. Εμείς το σκεφτόμαστε διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει τα γεγονότα, τις ε, προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην υγεία, στην ε, παιδεία, το θέμα των ανισοτήτων. Όλα αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε στην έκθεσή μας και να αναφέρουμε και τις ανησυχίε μας για τι εξελίξεις. Γιατί κατ' κατευθείαν επιδιώκουμε την οικονομική ανάκαμψη ε, των εν λόγω χωρών και αυτήν όμως την ανάκαμψη την καθιστούμε πιο δύσκολη εάν δεν αλλάξουμε ριζικά την εφαρμοζόμενη πολιτική. Άρα δηλαδή είναι αδιαμφισβήτο γεγονός ότι έχουμε αποφύγει τη διάλυση της Ευρωζώνης σε μία περίπτωση ε, παρεμποδίσαμε την άτακτη χρεοκοπία ενός κράτους μέλους. Βεβαίως γεγονός είναι αυτό και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναφέρουμε τα γεγονότα. Όμως από τη στιγμή που αναφέρουμε γεγονότα θα πρέπει να μην αναφέρουμε μόνο τα γεγονότα που αρέσουν ίσως σε κάποιους και δεν αρέσουν σε κάποιους άλλους. Όταν λοιπόν παραθέτουμε γεγονότα θα πρέπει να είμαστε όσο πιο περιεκτικοί γίνεται ακόμα και αν τα γεγονότα αυτά ε, περιλαμβάνουν, περικλείουν δυσάρεστες αλήθειες όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Τρόικα. Θεωρώ λοιπόν, αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, κατόπιν όσον αφορά τις πολιτικές συνέπειες ή τα συμπεράσματα του καθενό μας από τα γεγονότα, προφανώς και θα πρέπει να παραμείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στα στοιχεία που μας ενώνουν στην έκθεση και κατά τα άλλα νομίζω ότι κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να κάνει με αυτή την έκθεση ό,τι θέλει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Αυτές τις παρατηρήσεις ήθελα να κάνω αλλά και να επισημάνω το γεγονός ότι αν τελικά επιθυμούμε να υποβάλουμε ουσιαστικές προτάσεις στα όργανα, σε θεσμικό επίπεδο, θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους και να συμπεριλάβουμε όχι μόνο το κομμάτι εκείνο που έχει σχέση με την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης, αλλά και τη δική μας άποψη, που δηλαδή κατά την άποψή μας υπήρξαν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου ή για να το πω αλλιώς ποιες πολιτικές της ε, Τρόικα ήταν εκείνες που δεν ήταν νόμιμες και δεν εντάσσονται μέσα σε ένα ενωσιακό πλαίσιο. Και αυτό ήθελα να το θέσω επιτάπητος. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο σήμερα, αλλά θέλω να πω, κατά την άποψή μου, νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούν, εξ όσων γνωρίζω, ότι αυτή η διερευνητική έκθεση συντάχθηκε καθυστερημένα και πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά εφόσον επιθυμούμε να καταλήξουμε σε πολιτική κρίση και πολιτικές προτάσεις. Κάτω από αυτό το πρίσμα, εγώ θεωρώ, θα πρέπει ε, στην επόμενη θητεία να υπάρχει μια καλύτερα επανδρομένη, μια πλήρης ε, διερευνητική επιτροπή για το θέμα της Τρόικα. Επίσης, ελπίζω να επιτύχουμε ευρεία συμφωνία. Ξέρετε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να εξηγήσω γιατί οι πράσινοι διαφέρουν τις απόψεις τους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος. Ε, θέλω η όλη διαδικασία να είναι συμμετοχική, να συμμετέχουμε όλοι μας, αλλά να καταλήξουμε και κάπου, να προκύψει ουσία. Δεν θέλω δηλαδή αυτή να είναι μία έκθεση όπου να ε, προκύψουν πολιτιστικοί διαξυφισμοί μεταξύ ημών. Για το ECR δεν φαίνεται εδώ ο εκπρόσωπός τους. Για την ΚΟΕ. Γιούργεν. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, γιατί για μένα τουλάχιστον αυτό ήταν το πιο, η πιο σημαντική αποστολή που έζησα στη διάρκεια της θητείας μου. Και κατά όψι μας, το είπε και ο Φίλιπ αυτό, όλα αυτά που ακούσαμε ήταν πολύ σημαντικά γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να διαβάζει κανείς κάτι, να ακούει κάτι και να το βλέπει επιτόπου από τους ανθρώπους που πλήττονται και αυτό οδήγησε στο ότι πολλοί από αυτούς που πλήττονται εξέφρασαν μία σειρά προσδοκιών στην Κύπρο σίγουρα, αλλά και στην Ελλάδα. Μας είπαν δηλαδή, ελπίζουν, ή να το πω αλλιώς, Καταρχήν ε, χάρηκαν πάρα πολύ που πήγαμε και μας είπαν «Α, επιτέλους έρχεται και κάποιος από τις Βρυξέλλες, δεν κάθεστε μόνο στις Βρυξέλλες και να μιλάτε εκεί, αλλά έρχεστε εδώ επιτόπου, επιτόπου και συζητάτε μαζί μας». Αυτό λοιπόν για πολλούς ε, πολίτες ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Παράλληλα όμως τους ε, ενέπνευσε την ελπίδα ότι όσον αφορά την επιδίνωση των κοινωνικών μέτρων, γιατί αυτό το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι έχουμε, βλέπουμε, βιώνουμε μια κοινωνική επιδίνωση, Εκεί λοιπόν στο θέμα το κοινωνικό άρχισαν να τρέφουν ελπίδες ότι κάτι θα γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι ως Κοινοβούλιο φέρουμε κάποια ευθύνη για το πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα. Και πρέπει να το θίξουμε στην έκθεση, να αναφέρουμε και τα συμπεράσματά μας από όλα αυτά που είδαμε. Δεν θέλω κι εγώ να φορτίσω την όλη υπόθεση ιδεολογικά. Συμφωνώ με τον κύριο Κάρας ότι δεν θα πρέπει αυτή την περίπτωση να τη μετατρέψουμε σε ιδεολογική αρένα, να εξετάσουμε ρεαλιστικά τα προβλήματα, αλλά θέλω να υπογραμμίσω και αυτό που είπε ο Φίλιπ. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι με κάθε τίμημα να καταλήξουμε σε μια ανούσια έκθεση. Αυτό δεν θα κανένα, ούτε και εμά ω Κοινοβούλιο. Και συμβαστικές ε, τροπολογίες του Λίαμ και του Ότμαρ. Τελικά καταλήγω στο ότι πράγματι θα καταλήξουμε, ε, θα παρουσιάσουμε μια καλή έκθεση. Δηλαδή ε, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλοι με τις απόψεις, νομίζω αυτό είναι απόλυτα σαφές. Τώρα, όσον αφορά εμένα, θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα που με εντυπωσίασαν. Καταρχήν είναι όπως σας είπα η επιδίνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό το είπε ο Νίλ ε, και αυτό με εντυπωσίασε και εμένα γιατί αφορά συγκεκριμένα ανθρώπου. Στην Ελλάδα το είδαμε αυτό. Είδαμε την επιδείνωση του ε, συστήματος υγείας από τα περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους Ελλάδας, πάνω από 3 εκατομμύρια αποκλείονται, έχουν περιθωριοποιηθεί από το κοινωνικό σύστημα. Και όπως μας είπαν και πολλοί γιατροί, υπήρξαν αρκετοί θάνατοι όπου θα μπορούσαν αυτοί να έχουν αποφευθεί εάν οι άνθρωποι είχαν τύχει σωστής πρόνοιας και μεταχείρισης. Βέρνερ, αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει κανείς να την δει. Ξέρω ότι αυτό δεν το ακούν ευχάριστα οι Γερμανοί, αλλά συνέβη αυτό. Πρέπει κανείς να το έχει κατά νου. Αυτό λοιπόν είναι η κοινωνική επιδείνωση. Αλλά και σε πολιτικό επίπεδο αποκόμισα την εντύπωση ότι στις τρεις μικρές τουλάχιστον χώρες, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, το αίσθημα που επικρατεί είναι ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά η δυνατότητα να εκφράσουν οι χώρες αυτές την άποψή τους. Ότι δηλαδή υπήρξε μία ανισορροπία δυνάμεων από τη μια η ευρωομάδα και από την άλλη κάποιες μικρές χώρες οι οποίες δέχτηκαν αφόρητη πίεση από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Εγώ λοιπόν για καθαρά πολιτικούς λόγους αυτό το θεωρώ απαράδεικτο, ότι μικρές χώρες ε, να βρίσκονται σε τόσο μεγάλη κάτω από τόσο μεγάλη πίεση. Στην Κύπρο μας είπαν, είχαν ε, την αίσθηση ότι τους είχαν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο. Και ο Λίαμ το ανέφερε αυτό σε κάποιες συνδέξεις που έδωσε. Αυτό λοιπόν το θεωρώ πολύ σοβαρό και σε μια ένωση όπως αυτή που επιδιώκει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνεται αποδεκτό. Αυτές είναι δύο-τρεις εντυπώσεις που αποκόμισα που όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικές για μένα και γι' αυτό το λόγο έκρινα ότι ήθελα να σας τις πω. Όσον αφορά τώρα στις ε, τροπολογίες που καταθέσαμε. Οι τροπολογίες αυτές ε, ακολουθούν δύο κατευθύνσεις. Η μία, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, η μία λοιπόν είναι ότι λόγω του απροσδόκητου της κρίσης και λόγω του ότι η κρίση έπληξε την Ευρωζώνη απροσδόκητα, τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αντιδράσει αμελητή, όταν όμως δεν έχει ε, στη διάθεσή του απαραίτητα εργαλεία. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι κατά πόσον υπάρχουν ε, οι ευρωπαϊκές συνθήκες, ε, το νομικό πλαίσιο που να αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, άρα δηλαδή τίθεται και το ερώτημα κατά πόσον μια τέτοια έκτακτη περίπτωση νομιμοποιεί την κατάφορη παραβίαση δικαιωμάτων ή, να το πω αλλιώς, κατά πόσον δικαιολογεί το μη σεβασμό κάποιων δικαιωμάτων. Σε κάποιες λοιπόν από τις ε, τροπολογίες μου εξετάζω ακριβώς αυτό το θέμα. Ε, ανατέθηκε ε, στην Αυστρία κάποια μελέτη αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης να εκπονήσει και αυτό μια μελέτη και αυτές τις δύο μελέτες τις ε, αναφέρω στις τροπολογίες μου. Η άλλη κατεύθυνση κατά την άποψή μου είναι η εξής όσο απαραίτητε και είναι οι μεταρρυθμίσεις και αυτό το στηρίζω εγώ επουδενή δεν ισχυρίζομαι ότι οι μεταρρυθμίσει ήταν περιτές σε αυτά τα κράτη. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι επ' αυτού συμφωνούμε όλοι μας. Γιατί αν δει κανεί σε αυτές τις χώρες, προφανώς και ήταν απαραίτητο να λάβουν χώρα μεταρρυθμίσεις. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον αυτές οι τέσσερις σχετικά μικρές χώρες της Ευρωζώνης, κατά πόσον οι χώρες αυτές με τις μεταρρυθμίσεις μπόρεσαν πραγματικά να επιτύχουν τη σταθεροποίηση του ευρώ. Ή μήπως η ευρωκρίση ήταν εκείνη η οποία προήλθε από το ίδιο το ευρώ, από τον τρόπο δόμησης του ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να αποφύγουμε αυτό το ερώτημα το οποίο μπορεί να δυσαρεστεί τις μεγάλες χώρες αλλά παρόλα αυτά πρέπει να διερωτηθούμε τι ρόλο παίζει η διάρθρωση της Ευρωζώνης. Γιατί αν δεν το υποβάλουμε αυτό το ερώτημα, μετά από δύο-τρία χρόνια θα διαπιστώσουμε ότι αυτά τα οποία κάναμε κατ' ουσίαν δεν οδήγησαν πουθενά. Τώρα, και κάτι άλλο που το είπε ο Ότμαρ. Να αναζητήσουμε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Αυτή η πρόταση κατατέθηκε τουλάχιστον στη Γερμανία όταν ξέσπασε η κρίση και τη στηρίζω αυτή την πρόταση. Βεβαίως σε τελική ανάλυση το θέμα δεν είναι πώς ακριβώς θα πρικοδοτηθεί ένα τέτοιο ταμείο. Ε, η ιδέα βέβαια για μένα είναι πολύ σημαντική να υπάρξει ένα τέτοιο ευρωπαϊκό ταμείο και με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουμε το δρόμο προς ενωσιακές μεθόδους. Ε, στο σημείο αυτό, Βέρνερ, επειδή παρίστασε, θέλω να πω το εξής. Νομίζω κατά την άποψή μου στη Γερμανία οι αντιδράσεις του τύπου ήταν πολύ σκληρές σε κάποια στοιχεία της αποστολής μας. Μερικοί ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει κανένα δημοκρατικό έλλειμμα. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Η ισχυρότερη χώρα και ελέγχθη αυτό επανειλημμένα. Το είπαν συνάδελφοι από την Κύπρο. Είπαν επανειλημμένα ότι η Γερμανία έχει πάρει όμοιρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Καθαρά πολιτικά όμως το βρίσκω ολέτριο να προκαλείται αυτή η εντύπωση. Και νομίζω και ότι είναι προς όφελος της Γερμανίας να αποστρέψει αυτή την εικόνα, να μην παραμείνει η εικόνα αυτή προσκολλημένη στη Γερμανία, ότι δηλαδή η Γερμανία είναι η μόνη χώρα η οποία θέλει να καθορίζει τα πάντα. Ε, και νομίζω ότι Πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό, Βέρνερ. Ε, ποτέ δεν ήταν η θέση της Τσεντεού των Δημοκρατών ότι η Γερμανία θέλει να διαδραματίσει αυτό το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι ως Γερμανία πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας, το πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την εικόνα ε, και γενικότερα και κάποιες συμπεριφορές που νομίζω ότι είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Ο Λίαμ ρώτησε ε, και κλείνω με αυτό κατά πόσον επαρκεί το χρονικό διάστημα. Εγώ ελπίζω πως ναι θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε μια λογική έκθεση, σε λογικές συμβαστικές προτάσεις, να ολοκληρωθεί η έκθεση. Βεβαίως και δεν μπορούμε την έκθεση αυτή να την παραδώσουμε στο επόμενο κοινοβούλιο. Εμείς κάναμε την, εμεί συμμετείχαμε στην αποστολή και εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να ολοκληρώσουμε την έκθεση, όχι το επόμενο κοινοβούλιο και αυτή η έκθεση θέλω να πιστεύω ότι θα είναι το σημείο εκκίνησης, το εναρκτήριο λάκτισμα για περαιτέρω εργασίες. Αυτά εκ μέρους μου και ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Για να δω τώρα ποιοι ζήτησαν το λόγο. anybody else? Τελευταίος ο κύριος Χουντής, κανείς άλλος. Κυρία Κράτσα. Όλε. Άλλος. και εγώ, κι εγώ, κι εγώ η ίδια. Μάλιστα και εσείς κυρία Παπαδοπούλου. Όχι, εγώ θα μιλήσω τώρα γιατί θέλω να απαντήσω σε μερικά από αυτά που τέθηκαν. Δυστυχώς από μερικούς που έφυγαν ήδη. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε γιατί κάνουμε αυτή την έκθεση της Τρόικα. of uh, the Troika and, its actions. Uh, και γιατί αποφασίσαμε να αξιολογήσουμε την Τρόικα και τις δράσεις. Ο Φίλιπ Λάμπερτς έθεσε τις οικονομικές συνέπειες και τις υπόλοιπες συνέπειες. Προφανώς και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ευαίσθητοι εδώ. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε προς τα έξω, προς το κοινό, ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό και πέραν αυτού τίποτα. Αλλά πρέπει να δώσουμε κάποιες εξηγήσει γιατί κάνουμε τη συζήτηση αυτή πρέπει να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και για τον οικονομικό ευρύτερο κύκλο και για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην, στην ευρύτερη οικονομία και τι συνέπειες θα έχουμε μακροοικονομικά. Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Αν περάσουμε σε υπερβολικά επίπεδα θα έλεγα λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στο κοινωνικό τομέα, έχοντας σταθεί πρώτα βέβαια στις οικονομικές επιπτώσεις, τότε φοβάμαι ότι θα ε, τεθεί κάποιος ε, κίνδυνος σε σχέση με την ε, διείσδυσή μας στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. και θα πρέπει να προσέξουμε και τις διατυπώσεις έτσι ώστε οι προτάσεις μας να παραμείνουν στις αρμοδιότητές μας και όχι πέραν αυτών. Είναι επικίνδυνο το πεδίο αυτό, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παρετηθούμε μπροστά στο μέγεθος δυσκολίας αυτής της προσπάθειας για το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι αφού Ολοκληρώσαμε την έκθεση. Θέλουμε κάποιο χρόνο όσο είμαστε εδώ μαζί για να μπορέσουμε να την διαμορφώσουμε έτσι ώστε να την παρουσιάσουμε. δεν θα πρέπει εμείς να τελειώσουμε την τελευταία στιγμή τη διαδικασία και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να πει ό,τι θέλει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Θα πρέπει όσο είμαστε μαζί εδώ όσο συνεδριάζουμε σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο, να σταθούμε ικανοί να ε, προβάλλουμε προς τα μέσα ενημέρωση την συλλογική μας άποψη, τη συλλογική μας εικόνα. Κάτι το οποίο θα δείξει το επίπεδο ευθύνης μας. Λοιπόν, δεν θέλω ε, κάποια σχόλια ακόμα για να μην σας ενοχλήσω εκ νέου. Θα αναφερθώ σε πέντε δικές μου τροπολογίες, λίγες είναι. Τρία θέματα να υπογραμμίσω. Το πρώτο, στην 831, ε, δείχνει το πώς στρατηγικά η σκέψη γύρω από το Μπέιλιν εξελίχθηκε με το χρονο was not an um, Είδαμε πώς εφαρμόστηκε αυτό στην Κύπρο, όπου τέθηκε το θέμα των καταθέσεων βέβαια. και συνολικά του κόστους. γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει στην Ελλάδα. Νομίζω λοιπόν ότι και στα πλαίσια της πρότασης τώρα για την οδηγία για την... And, and σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονται για την οδηγία για το κλείσιμο των τραπεζών, για την εκαθάριση εν πάση περιπτώσει των τραπεζών προτείνονται συγκεκριμένα ποσοστά και πράγματι θα πρέπει να δούμε μικρές χώρες να μην αναλαμβάνουν υπερβολικά, υπερβολικά βάρη προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Πράγματι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργούμε σαν transfer union, σαν υπηρεσία μεταφοράς ε, ποσών δεξιά και αριστερά, αλλά στην προσπάθεια διάσωσης των οικονομιών πράγματι έγιναν κάποιες τέτοιες προτάσεις. Στα πλαίσια της 829 και της 832 δείχνω ακριβώς την ευελιξία που είναι διαθέσιμη στο Σύμφωνο για την Ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο κάναμε και στο διπλό πακέτο προτάσεων. Νομίζω ότι αργότερα θα πρέπει εμείς να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα και τις δυνατότητες άμεσης ανακεφαλαιοποίησης από τον ESM. Αυτά όμως για το μέλλον. Θέματα τα οποία προσπάθησα να θίξω με κάποια ευαισθησία. Υπάρχουν θέματα δικαιοσύνης εδώ για το τι στην ουσία συνιστά μεταφορές προς όφελος των χωρών που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Για την 390 που κατέθεσα εκ των υστέρων, ανησύχησα για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδα και στα μέσα ενημέρωση το τι συμβαίνει στην παρούσα φάση στην Κύπρο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς βέβαια στο βάθος των υποθέσεων αυτών χωρίς να κάνει τις απαιτούμενες έρευνες. Είχαμε και κάποιες αντίστοιχες καταστάσεις, ίσως όχι τόσο οξυμένες και στην Ισπανία, όπου υπήρξε μια αλλαγή κυβέρνησης και αμέσως μετά ακολούθησε και η αλλαγή του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ξέρω αν τέτοιου είδους μέτρα είναι τα πιο κατάλληλα και πρέπει να συμβαίνουν, όταν σύμφωνα με τη συνθήκη είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ανεξάρτητους κεντρικούς τραπεζίτες. Εγώ τα αναφέρω αυτά στην τροπολογία μου με πολύ συγκεκριμένο ε, τρόπο. Ε, κοιτάξτε, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Λίγη ησυχία παρακαλώ, γιατί δεν, δεν ακούω τι, τι λέω όταν εσείς μιλάτε. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι ε, πολύ ενδιαφέρον. Επηρεάζει και τον ρόλο της Τρόικα και τον ρόλο ε, των κεντρικών τραπεζών που έπαιξαν σε σχέση με τις κατεπίγουσες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στον τομέα της ρευστότητα, σαν παράδειγμα των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα και πολλές φορές οι αποφάσεις τις οποίες έλαβαν ήταν καρπός υπερβολικής πίεσης. Πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προβλήματα σε σχέση με την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Είναι θέματα αυτά τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε ε, και χωρισμένα, θα έλεγα σε μια ιστερότερη φάση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. <coughs> Διόγκο. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους εκείνους ε, οι οποίοι συμμετείχαν ε, σε αυτή την εκπόνηση της έκθεσης. Και διότι σε τελική ανάλυση αυτά που μας υποβλήθησαν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κάρας Ευχαριστώ τον κύριο Κάρας για την ε, βοήθειά του, γιατί οτιδήποτε μας είπε βασίζεται στην κοινή λογική, στον κοινό νου, σε όλες του τις ε, δημόσιες ε, δηλώσεις δεν προέβη καμία φορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, που δεν προκάλεσε ποτέ, ποτέ δεν ε, θέλησε να διαιρέσει την ομάδα και γι' αυτό λοιπόν τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Συμφωνώ μαζί του ότι χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την έκθεση. Δεν χρειαζόμαστε επουδενή την ε, ιδεολογικοποίηση της συζήτησης γιατί αυτό θα οδηγούσε σε διέρεση της ομάδας. Θα ήταν σαν να διεξάγουμε πρόωρα προεκλογική εκστρατεία, κάτι που δεν θα ωφελούσε κανέναν τελικά. Και θέλω να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι τελικά είμαι σίγουρος θα έχουμε μια έκθεση η οποία θα συγκεντρώσει την μέγιστη δυνατή πλειοψηφία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να παραμείνουμε μέσα σε κάποια όρια της συζήτησης. Δεν πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα για το πρόγραμμα ΑΒΓ της ΑΒΓ χώρας, αλλά να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είδους συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε για το μέλλον. Εάν λοιπόν παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο, τότε για μένα θεωρώ ότι θα έχουμε πράξει το σωστό. Και το τονίζω αυτό γιατί εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Πορτογαλία, η οποία εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα προσαρμογής και παρόλα αυτά σας λέω δεν έχει κανένα νόημα να αρχίσουμε τη συζήτηση για το ποιος τελικά επέβαλε ποιο πρόγραμμα σε ποια συγκεκριμένη χώρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τελικά αυτό δεν παίζει μεγάλο ρόλο για μας. Βεβαίως συνέβησαν πράγματα τα οποία ποτέ δεν έπρεπε να λάβουν χώρα στα κράτη-μέλη θα έπρεπε ίσως ε, να έχει δοθεί η απάντηση πολύ νωρίτερα, αλλά επίσης όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το να υπάρχει απόλυτη αδράνεια, αυτό δεν είναι λύση. Σίγουρα υπήρξαν πράγματα που έκανε η Τρόικα, που ήταν ε, λάθος, ε, αλλά υπήρξαν και άλλα που ήταν σωστά. Ε, ε, που δεν είδε πρέπει να καταληγεί κανείς το ότι η Ευρώπη δεν έπρεπε να κάνει τίποτα και να παραμείνει αντρανής. Τώρα χρειαζόμαστε μια σταθερή στάση που να βασίζεται σε ενωσιακές πρακτικές. Οτιδήποτε άλλο δεν θα βοηθήσει. Δεν θέλω να σπαταλίσω το χρόνο σας και γι' αυτό ολοκληρώνω λέγοντας ότι έχω καταθέσει Μία τροπολογία που παρακαλώ να τη λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τους οι συγητές είναι η τροπολογία εκείνη που περιγράφει την κατάσταση των τεσσάρων κρατών μελών που βρίσκονται σε πρόγραμμα όταν ξεκίνησε και ξέσπασε η κρίση. Σε τρία από τα κράτη-μέλη τα οικονομικά δεδομένα αφορούν το έτος πριν από την εφαρμογή του προγράμματος. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τα στοιχεία της Πορτογαλίας προέρχονται και αφορούν το 2007 όταν ακόμα δεν είχε ξεσπάσει η κρίση. Εχθές λοιπόν προσπάθησα να δω μόνος μου ε, τι ακριβώς έγινε το 2007 στην Πορτογαλία και από πού προήλθαν αυτά τα στοιχεία και τελικά ήταν η ημερομηνία, η χρονιά εκείνη όπου υπογράφηκε η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, ήταν η χρονιά επίσης ε, που είχαμε το διεθνές έτος ε, του Δελφινιού αλλά κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν τα βρίσκω σημαντικά για να τα λάβουμε ως ε, έτος αναφοράς για την Πορτογαλία. Με συγχωρείτε, αλλά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι τα ίδια για όλες τις χώρες διότι θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος της Πορτογαλίας. Εγώ έχω καταθέσει τροπολογία που να λέει ότι τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι από την ίδια χρονιά για όλες τις χώρες όταν δηλαδή ξέσπασε η κρίση. Και δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους συνεισηγητές. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Sharon για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Διέγκο. Ε, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να υπογραμμίσω ότι αυτή η επιλογή, η επιλογή της συγκρότησης των Τρόικα σε πρώτη φάση στην Ελλάδα και ακολούθως στα υπόλοιπα κράτη-μέλη ήταν μια αναπόφευκτη επιλογή με τα δεδομένα εκείνης της περίοδου για να αποτραπεί και να αποφευθεί ελλείψη οποιονδήποτε μηχανισμών και πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης εκείνη την περίοδο, μία άτακτη χρεοκοπία με συνέπειες πολύ δυσμενέστερες από αυτές που υπέστησαν οι χώρες σε πρόγραμμα και η Ευρωζώνη συνολικά. Ε, θέλω με τη σειρά μου να πω αυτό που υπογράμμισαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι αυτό το εγχείρημα της σύνταξης αυτής της έκθεσης διερεύνησης είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, ήταν και είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, οι δύο συνεισηγητές, ο ε, Ότμαρ Κάρας και ο Λίεμ Γκότς, δεν αξίζουν μόνο ευχαριστίες, πιστεύω ότι αξίζεται συγχαρητήρια γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο και παραμένει μέχρι τέλους πολύ δύσκολο να κατορθώσετε να γεφυρώσετε τις διαφορετικές απόψεις μέσα στο κοινοβούλιο γύρω από ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και να δημιουργήσετε μία σύνθεση και κάποιους, ε, κάποιες ε, συμβιβαστικές προσεγγίσεις που ταυτοχρόνως έχουν περιεχόμενο και αυτό αντικατοπτρίζεται στις συμβιβαστικές προτάσεις που έχετε μέχρι σήμερα. Πιστεύω και εγώ, όπως είπε και ο Γιούργεν και ο Φίλιπ, ότι για το Κοινοβούλιο έχει πολύ μεγάλη σημασία, παρά το γεγονός ότι η έκθεση αυτή δεν ε, πρέπει να είναι εργαλείο προεκλογικής καμπάνιας οποιοδήποτε κόμματος, πιστεύω όμως ότι έχει μεγάλη σημασία για την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου, απευθείας εκλεγμένου από τους πολίτες, ελάχιστο διάστημα πριν από τις ευρωεκλογέ, το τελικό αποτέλεσμα που θα επικυρωθεί βεβαίως από την Ολομέλεια. Εύχομαι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία να είναι τεκμηριωμένο, ισορροπημένο, περιεκτικό και να αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις και στρατηγικές προσεγγίσεις του Κοινοβουλίου ε, συνολικά, ε, κυρίως για το μέλλον, για το επόμενο διάστημα. Και συμφωνώ, Ότμαρ, ε, το υπογράμμισαν και άλλοι ομιλητέ ότι για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις ε, ιδεολογικές προσεγγίσεις. Ε, δεν πρέπει να είναι αυτές οι κυρίαρχε, γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ποτέ σύνθεση. Όμως πρέπει ταυτοχρόνω να έχουμε υπόψη ότι οι συζητήσει μας και το τελικό μα αποτέλεσμα παρακολουθείται από του πολίτε κυρίω των χωρών που εφαρμόζουν πρόγραμμα. Σωστά είπε ο Φίλιπ ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να εκπέμπει το μήνυμα ότι ασχολείται μόνο με τους αριθμούς, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Και το επισημαίνω για να πω το εξή ότι όπως εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει οι ιδεολογικοκεντρικές προσεγγίσεις να ε, μένουν ε, στην άκρη, αυτό το μήνυμα θεωρώ ότι πρέπει να το εκπέμπουμε ως Κοινοβούλιο και να το εκπέμψουμε και με την τελική μας έκθεση, και προς τις τρόικες στις χώρες που εφαρμόζουν πρόγραμμα προσαρμογής. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί εμείς σήμερα συζητάμε, αλλά υπάρχουν χώρες όπως η δική μου ε, που βρίσκονται σε μια φάση μίας ακόμη πολύ δύσκολης αξιολόγησης και θέλω να σας δώσω ως παράδειγμα ότι στο πλαίσιο αυτής της πολύ δύσκολης αξιολόγησης, αυτές τις μέρες που εμείς συζητάμε εδώ, η Τρόικα ζητάει από τις ελληνικές αρχές να θεσπίσει ένα νόμο που απελευθερώνει τις μαζικές απολύσεις. Και λέω λοιπόν ότι σε μια χώρα που έχει 28% ανεργία, βρίσκεται στον έκτο χρόνο της ύφεση, που βρίσκεται σε αποπληθωρισμό, δεν είναι σε κίνδυνο αποπληθωρισμού, ως συνέπεια του ραγδαίου αποπληθωρισμού των μισθών, Υπάρχει ήδη αποπληθωρισμός που περιπλέκει τη βιωσιμότητα του χρέους στην Ελλάδα. Και λέω αυτού του είδους οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι που πρέπει να έχουν προτεραιότητα σήμερα σε μια χώρα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το one fit for all λοιπόν που παραπέμπει σε ιδεολογικά στερεότυπα πρέπει να το καυτηριάζουμε γιατί ακριβώς όπως έλεγα και πριν μας παρακολουθούν ε, οι πολίτες κυρίως των χωρών που έχουν οικονομικές δυσκολίες, τις συζητήσεις μας και το τελικό μας αποτέλεσμα. Σε σχέση με τις τροπολογίες, πολύ σύντομα, ε, θέλω να πω καταρχήν ότι συμφωνώ απολύτως με τον Ότμαρ ε, στην ε, προτεραιότητα που έδωσε στο ζήτημα της κοινοτικής μεθόδου και της κοινοτικής νομοθεσίας και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό αντικατοπτρίζεται στην έκθεση ε, ήθελα μόνο να επισημάνω ότι στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης έχω υποβάλει ε, μια τροπολογία, την τροπολογία 133, που επισημαίνει, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία με την κουβέντα που κάνουμε σήμερα, ότι ε, βραχυπρόθεσμα η χορήγηση οικονομικής βοήθειας στόχευε ασφαλώς την αποτροπή της άτακτης χρεοκοπίας, μέσω μακροπρόθεσμα δεν θεωρώ σωστό να λέμε ότι η χορήγηση οικονομικής βοήθειας στοχεύει στην αποπληρωμή των δανείων ώστε να μην επομιστούν το βάρος οι φορολογούμενοι των άλλων χωρών. Είναι αυτονόητο ότι ε, ε στόχος μας είναι η αποπληρωμή των δανείων, στόχος μας είναι να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι των άλλων χωρών, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί και αυτό επιδιώκουμε εμείς ε, μέσω ε, τις ε, ε, βοήθειες που δίνουμε στις οικονομίες των χωρών αυτών να ξανασταθούν στα πόδια τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Επίσης, ένα άλλο σημείο υπογραμμίστηκε και από άλλους συναδέλφους που νομίζω ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων και πρέπει να υπογραμμιστεί από το Κοινοβούλιο η ανάγκη συμβατότητας και η κριτική όπου δεν υπήρξε αυτή η συμβατότητα των προγραμμάτων με την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει σε αυτό το θέμα που είναι στρατηγικό για μας ε, να, ε, να μην είναι πολύ αυστηρό. Και τέλος, μία παρατήρηση μόνο σε ό,τι αφορά τις, τις αναφορές στη χώρα μου, στην Ελλάδα. Ε, εγώ, όπως ξέρετε, γιατί γνωριζόμαστε πια πολλά χρόνια, ε, είμαι ο τελευταίος που θα αρνούμουν την κριτική στη χώρα μου και για τις ευθύνες που οδήγησαν στην κρίση αλλά και κριτική που έχει να κάνει με καθυστερήσεις, με ελλείψεις στην εφαρμογή. Όμως θα θεωρούσα άδικο να μην επισημάνουμε και η σχετική παράγραφος ε, στο, ε, στην, στο draft report εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη πρόοδου στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι άδικο στην ελλάδα έχει σημειωθεί μια δημοσιονομική προσαρμογή άνευ προηγουμένου ε, ε, εξαιτίας θυσιών των ελλήνων πολιτών που δεν επιμερίστηκαν και με το δικαιότερο τρόπο όπως ξέρουμε και νομίζω ότι και αυτοί οι πολίτες αλλά και οι πολίτες των υπόλοιπων χωρών που τους βοήθησαν αξίζουν αυτή την αναγνώριση δηλαδή ότι υπάρχει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι τα προγράμματα ήταν δύσκολα στις περισσότερες χώρες με την έννοια ότι μεταρρυθμίσεις που για ολόκληρες δεκαετίες δεν είχαν εφαρμοστεί έπρεπε να εφαρμοστούν ε, βία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό συνέβη στα κράτη-μέλη, βέβαια με κάποιες διαφορές. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων σε όλους αυτούς που λένε ότι η προσέγγιση πρέπει να στερείται η ιδεολογική τοποθέτηση. Η όλη η τοποθέτηση ε, για την έκθεση δεν ήταν ιδεολογικά φορτισμένη. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με τις τροπολογίες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι Πολλοί είπαν ότι δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Τομείο. Κοιτάξτε, αυτό τι δεν είναι απέναντί μας υπόλογη και αυτό όμως αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το επέτρεψε αυτό και σε πολλά άλλα κράτη και στη Γερμανία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν έχει πολύ μεγάλη εξουσία στην κοινή αγορά. Υπολείπεται κατά πολύ το επιθυμητού και εγώ συμφωνώ με όλους εκείνους που το επικρίνουν αλλά δεν ξέρω πόσο υψηλός ε, είναι ο κίνδυνος ε, να παραπεμφθεί κανείς ε, για μη τήρηση των συνθήκων. Ξέρετε και η Γερμανία παραπέμπεται και έχει παραπεμφθεί επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τέτοια ε, για διαδικασίες επί παραλήψη. Στη δεύτερη θέση βέβαια έρχεται η Ελλάδα και στην τρίτη θέση είναι η Γαλλία. Κατόπιν τούτου αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε απαραίτητα να κάνουμε μεγάλα μικρά μεσαία κράτη. Έχουμε να κάνουμε, θα το πω ως εξής. Έχουμε να κάνουμε με παρατηρήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 10 ολόκληρα χρόνια που δεν παρενέβη, που δεν έκανε απολύτω τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξή. Το αίτημα να υπάρχει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο και η Τρόικα ε, να είναι μόνο μία έκτακτη περίπτωση, αυτό εγώ δεν συμφωνώ. Η κυρία Ποδηματά είπε ότι τότε δεν υπήρχε άλλη λύση και εγώ συμφωνώ επ' αυτού. Τότε δεν υπήρχαν άλλα εργαλεία δεν υπήρχαν μοντέλα, πρότυπα να εφαρμοστούν. Μπορεί κανείς να διαφωνεί για τα μακροοικονομικά πρότυπα. Και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά ξέρετε, όλα τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, στη τελική ανάλυση συζητήθηκαν ενδελεχέστατα με τα κράτη-μέλη, αποφασίστηκαν και στην περίπτωση της Κύπρου, εκεί υπήρξε πράγματι ένα τύχημα. Το εξή, η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε να συμπεριληφθούν οι καταθέσεις των ιδιωτών. Αυτό ήταν ένα αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης που αναθεώρησε μετά από μία εβδομάδα. Δεν ήταν αίτημα της Τρόικα, ήταν αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης. Και να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Και η διαφορά μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας είναι πρόδειλη. Δηλαδή, στην Ελλάδα, δεν θα υπερβάλλω, η Άννη μόλις τώρα αναφέρθηκε στην τροπολογία μου 226 για την οποία είχε παραπονηθεί σε μένα έτσι και αλλιώς και η κυρία Κράτσα. Το θέμα είναι ότι δεν αρκούν ε, οι αποφάσεις αν δεν εφαρμόζονται. Ε, στις άλλες χώρες τα πράγματα ήταν ε, καλύτερα από ό,τι συνέβη στην Ελλάδα. Λυπάμαι πολύ. Εντάξει, αν θέλετε μπορούμε να διαφωνήσουμε για τη διατύπωση, αλλά αν θέλετε να έχουμε μια καλή έκθεση θα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά την Πορτογαλία, αν ισχύει αυτό που ελέγχει ότι οι χώρες εδέχτησαν αφόρητη πίεση, ε, τότε αυτό ισχύει μόνο για την Πορτογαλία. Όλα τα άλλα οι χώρες τα προκάλεσαν μόνες τους. Πράγματι, στην Πορτογαλία η Κομισιόν και ο πρόεδρος Μπαρόζο άσκησαν αφόρητη πίεση να μπει η Πορτογαλία υπό την προστατευτική ασπίδα. Δεν το ήθελαν αυτό οι Πορτογάλοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε πίεση. Γι' αυτό λοιπόν να μετακυλεί κανείς ε, την ευθύνη προς την Τρόικα, αυτό ε, δεν είναι σωστό. Να πω επίσης το εξής. Εγώ, ξέρετε, ήμουνα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν μιλάγαμε από το 1994 για την εφαρμογή προγραμμάτων σταθερότητας. Ξέρω πάρα πολύ καλά τη συνθήκη σταθερότητας και ξέρω πολύ καλά ότι η Ελλάδα το 2000 ε, κατέθεσε μια συμπληρωματική αίτηση, όπως εντωμεταξύ έχουμε μάθει σήμερα με βάση λάθος στοιχεία και εγώ τότε το 2000 δήλωσα αποχή στην ψηφορία. Αποχή δήλωσα, γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Και το γεγονός ότι με βάση πολιτικές ε, διασυνδέσεις ε, προχώρησε η αίτηση της Ελλάδας να μπει στην Ευρωζώνη, αυτό μεταξύ το ξέρουν όλοι. Και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης πρώτες το παραβίασαν η Γερμανία και η Γαλλία, όχι η Ελλάδα κατά δύο συναπτά έτη. Και αφού το έκαναν αυτό, μετά το κατέστησαν πιο άκαμπτο, δηλαδή μη εφαρμόσιμο. Και εγώ στη Γερμανία το λέω αυτό κάθε φορά που μιλώ δημόσιο. Δηλαδή, όποιο κατηγορεί τι μικρέ χώρε ότι δεν εφαρμόζουν ή δεν εφαρμόσαν ε, το σύμφωνο σταθερότητα, να απευθυνθεί καλύτερα στου κυρίου Σρόιντερ και Φίσερ που τότε, το 2004-2005, συνεργάστηκαν με του Γάλλου και παραβίασαν το σύμφωνο και τότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλησε να τις επιπλήξει. Δεν ήταν τότε η Ελλάδα. Ήταν άλλες οι χώρες. Γι' αυτό λοιπόν όταν η πολιτική ελίτ δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει σωστά προγράμματα στις μεγάλες χώρες, τότε πώς νομιμοποιούμε θα αναζητήσουμε το ίδιο από τις μικρές χώρες. Ίσως πράγματι, ορισμένα πράγματα να έπρεπε να γίνουν διαφορετικά. Όμως ε, τελικά η συνέπεια είναι ότι όλα αυτά σύρθηκαν, υπήρξαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ η πέτεια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η έκθεση αν πραγματικά δεν χρησιμεύσει ως προεκλογικό ε, εργαλείο θα πρέπει η έκθεση αυτή να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σε ορισμένες χώρες υπήρξε ένδια θάρρους. Ένδια μέτρων για να εφαρμόσουν αυτό που έτσι κι αλλιώ ήξεραν. Το 2000 η Γερμανία ήταν ο ασθενή τη Ευρώπη και τότε η κυβέρνηση, της οποία εγώ δεν ήμουνα ε, μέλο, το κόμμα μου λέει δηλαδή, δεν ήταν στην κυβέρνηση, τότε το κόμμα, το κυβερνών κόμμα, ενάντια στη θέληση των υπολείπων μελών, ο Γκέρχαρτ Σρόντερ, ο σοσιαλιστής, έθεσε την ε, επανεκλογή του σε κίνδυνο και εφάρμοστε στο πρόγραμμα. Αυτό όμως δεν το βλέπω στην Ελλάδα να υπάρχει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα τζάκια που έρχονται και επανέρχονται και δεν δείχνουν την προθυμία να ακολουθήσουν αυτήν την τακτική. Και τώρα που μιλάμε ανοιχτά έχει εξαφανιστεί και η τηλεόραση του Κοινοβουλίου, κάτι που συμβαίνει συχνά, γιατί εγώ σας λέω ότι σαφώς και υπάρχει πολιτικό θεματολόγιο. Το βλέπετε, να έφυγε η τηλεόραση. Τώρα που ασκώ κριτική εξαφανίστηκε η τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, next... Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χουντής. Δυστυχώς ο κύριος Λάγκεν ομιλεί εκτός μικροφώνου. Ανακάλυψα ένα σημείο που συμφωνώ με τον κύριο Λάγκεν που φεύγει ότι και εγώ διαμαρτύρομαι που λείπει η τηλεόραση της Βουλής. Και εσύ. Ωραία. Αλλά με τη γενικότερη έννοια του όρου αγαπητοί συνάδελφοι, δηλαδή να ακούσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι κάνουμε εμείς εδώ, θέλω να σας πω το εξής επειδή και κατά την έκθεση και κατά τις τροπολογίες άκουσα δύο πράγματα από τους συναδέλφους. Δεν φτιάχνουμε ένα ιδεολογικό κείμενο, μάλιστα, και δεύτερο, να αποφύγουμε τον προεκλογικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Για τον προεκλογικό χαρακτήρα. Δεν ξαναθέτω το ερώτημα πώς φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε όμως κύριε Κάρας, δεν ξέρω αν γελάτε αν συμφωνείτε, να καταλήξουμε σε αυτή την έκθεση πριν κλείσει το κοινοβούλιο μόλις και λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Πείτε μου τι συμπέρασμα θα βγάλει ο άλλος. Μπορούσαμε να το κάνουμε πιο νωρίς. Εγώ λέω μπορούσαμε. Με αυτές τις προδιαγραφές. Με αυτές τις προδιαγραφές. Το δεύτερο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν περιμένουν. Μπορώ να το πω Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, ο ελληνικός λαός δεν περιμένει από την έκθεση που θα τελειώσουμε εμείς στο τέλος του Μάρτη να βγάλει συμπεράσματα και πολύ περισσότερο να του εξηγηθούν όσα βιώνει τέσσερα χρόνια. Τα έχει βγάλει τα συμπεράσματα. Και θα τα δείτε και στις ευρωεκλογές και σε άλλες χώρες. Εμείς όμως έχουμε μια υποκριτική στάση και θα σας πω γιατί όλες αυτές τις ανακατατάξεις που έχει φέρει και το μνημόνιο και η τρόικα σε διάφορε χώρε όχι μόνο στη δική μου τη χώρα εμείς μέσα στην έκθεση το χαρακτηρίζουμε ότι οι πολιτικές αντιστάσεις είναι ένα από τα εμπόδια για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Εμεί το αξιολογούμε έτσι. Τι κρίνεται και ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα που κρίνεται από την έκθεση. Γνωρίζοντας και γνωριζόμαστε πια δεν περιμένει ο άλλος να ακούσει τα συμπεράσματα. Τα έχει καταλάβει, τα έχει δει, τα βιώσει. Δεν χρειάζεται ίσως και περισσότερη εξήγηση. Εν πάση περιπτώσει να την κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Θέλω να σας πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς και που είναι μια άσκηση νομικού ελέγχου, μια άσκηση αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πολλούς λαούς και για το λαό της χώρας μας είναι βίωμα. Το βιώνει καθημερινά. Πού κρινόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι αν αυτά που θα αποτυπώσουμε σε αυτή την περιορισμένη έκθεση είναι αντίστοιχα των γεγονότων. Συμφωνώ. Και θα σα πω των γεγονότων. Όχι τη αξιολόγηση εμένα, του κυρίου, των άλλων συναδέλφων. Και το πολιτικό πρόβλημα που βρίσκεται. Αν εν ώψη ευρωεκλογών δοθεί το μήνυμα στου πολίτε ότι εμεί που ερχόμαστε εδώ δεν έχουμε ξεκοπεί από την εικόνα και τα προβλήματα των χωρών, δεν κάνουμε απλώ ασκήσει, αλλά έχουμε αίσθηση το τι έχει συμβεί και κατ' επέκταση είναι ένα πρόβλημα δημοκρατίας σε όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν με την έκθεσή μας πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το τι έχει γίνει. Οι τροπολογίες που κατέθεσα στηρίζονται σε γεγονότα. Σας τα αναφέρω για να μην ε, ή τουλάχιστον να διευκρινιστούν. Πρώτον, είχαμε κάνει ακρόαση, επειδή κοιτάω τον κύριο συνάδελφο από τη Φιλανδία, επειδή λέει ότι έχουμε καθυστερεί ή προεκλογικό χάρη, Ακρόαση τη Τρόικα, κύριε συνάδελφε, είχαμε κάνει και με συγχωρεί που αναφέρομαι σε σένα, δεν Στι 27 Μαρτίου του 2012. Ναι. Τότε, αν δεν το είχαμε καταλάβει από την αρχή, διακρίναμε τα προβλήματα νομιμότητας και τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων. πάω στην νομιμότητα. Κατά την έκθεση. Πού βρίσκεται το πρόβλημα. Έτσι όπως στήθηκε η Τρόικα παραδεχτήκαμε όλοι ότι δεν ήταν νόμιμη. Και δεν είναι νόμιμη. Αυτό το ξέραμε ή θα μπορούσαμε να το διαπιστώσουμε από την αρχή. Το δεύτερο. Ο ρόλος της Κομισιόν μέσα στην Τρόικα. Της Κομισιόν. Το όργανο το οποίο ελέγχουμε. Έχω επαν... πάρα πολλά ερωτήματα και απαντήσεις η Κομισιόν, η οποία είναι θεματοφύλακας του κοινοτικού δικαίου, αντί να περιφρουρεί το κοινοτικό δίκαιο, όχι καμιά ανατρεπτικές πολιτικές, με τα προγράμματα της Τρόικα το παραβίαζε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το παραβίαζε. Εγνωσμένα, ομολογημένα, έχω πολλές ερωτήσεις, και τίθεται θέμα τελικά, την Κομισιόν εμείς μπορούμε να λέξουμε. Έχει ευθύνη. Αφήστε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, μην σα πιάσω. Η Κομισιόν έχει ευθύνη. Ότι δεν λειτουργούσε ω υπερασπιστή τη κοινοτική νομοθεσία. Όχι τίποτα παραπάνω. Ούτε φιλικά προ τον ένα, ούτε φιλικά προ τον άλλο. Και αυτό είναι διαπιστωμένο πολλέ φορέ. Εδώ υπάρχει ευθύνη. Και επομένω μπορούμε να ελέγξουμε εμεί. Το άλλο που θέλω να σα πω για να μην σα κουράζω περισσότερο, υπάρχει λοιπόν στο σκέλο τη νομιμότητα να πούμε ορισμένα πράγματα με το όνομά του. Πάω στα προγράμματα για να, μην ε, ε, τελειώσω, για να μην... στη βάση αυτών που είπε και σέβομαι τις απόψεις του κ. Κάρας. Τα προγράμματα πώς θα τα αξιολογήσουμε. Δεν θα αναζητήσουμε την κοινωνική νομιμοποίηση. Αυτές οι καταστροφές έγιναν γενικώ, λέει κάπου και κάνω μια διαφορετική τροπολογία. Τα προγράμματα λέει, θα το πω αργά για να βοηθηθεί η μετάφραση, δεν δεσμεύονται από το χάρτη δεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι. Παραβίαζαν το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το έχουν ομολογήσει. Το έχουν διαπιστώσει και οι Κομισιόν πολλές φορές και άλλοι. Το έχουν πει. Τι πάει να πει δεν δεσμεύονται. Εάν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό τον... Έχουν παραβιάσει τα προγράμματα, έχουν παραβιάσει. Και μπορώ να σας αναφέρω αρκετά πράγματα, όπως και η περίπτωση που αναφέρθηκε η συναδέλφισσα για τις ομαδικές απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά τα προβλήματα. Κοινοτική νομοθεσία σας λέω, όχι κάποιο άλλο νομοθεσία. Έχουν παραβιαστεί. Και όσο αφορά τα αποτελέσματα, πολλές τροπολογίες αναφέρουν αποτελέσματα, στοιχεία. Δεν είναι από το κεφάλι μου που πρέπει να συμπληρωθούν. Ναι, τελειώνω, τελειώνω. Που πρέπει να συμπληρωθούν. Δεν είναι καμιά πολιτική αξιολόγηση είναι τα στοιχεία. Ότι φτάσαμε σε αυτό. Και έχει αξία, αγαπητοί συνάδελφοι, για να πάει η αξιολόγηση να δει κανένα τι θα κάνει, αφού καταγράψει την καταστροφή που έχει γίνει, αφού καταγράψει το αδιέξοδο, να πει κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Όχι να πει δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, μπορούσαμε, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, αλλά τώρα πρέπει να συνεχιστούν για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και τελειώνω. Σε αυτό εδώ ο πολιτικό πειρασμό μπήκε και στην επίσκεψη στην Ελλάδα. Το παρακάμπτω ως ένας ατυχές γεγονός, αλλά μην κάνουμε πως δεν χωράει πολιτική εκμετάλλευση το τι θα πει η έκθεση. Ξαναλέω, τα συμπεράσματα έχουν βγει, τη δική μας αξιοπιστία και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ας υπερασπιστούμε. Αυτές, αυτό είναι το πνεύμα των δικών μου τροπολογιών. Θα δούμε πώς θα πάει στα πράγματα. Τελείωσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Uh, Συγγνώμη που σας διακόπτω πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, αλλά έχουμε άλλους τρεις ομιλητές και θα ήθελα και οι συγητές να πάρουν το λόγο. Γι' αυτό παρακαλώ προσπαθήστε να είστε σύντομοι. Η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές για όλο το χρόνο και την ενέργεια που έχουν βάλει σε αυτή την υπόθεση τις επισκέψεις τους στις χώρες που είναι υπό πρόγραμμα ε, προσαρμογής στην Ελλάδα, στην Αθήνα παρακολούθησα και εγώ την επίσκεψή τους και είδα πραγματικά πόσο θέλανε να καταλάβουν όλες τις πλευρές των εξελίξεων ε, με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με όλα τα πολιτικά κόμματα όπως έγινε στο Εθνικό Κοινοβούλιο Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι ανεξάρτητα αν είμαστε ή όχι σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και υπεύθυνοι με αυτή την έκθεση. Διότι και οι πολίτες παρακολουθούν και, οι πολιτικοί παράγοντες σε όλες τις χώρες της Ένωσης, όχι μόνο στις χώρες που είναι με πρόγραμμα κανείς δεν μπορεί να φανταστεί και να υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε πολλές περιπτώσεις, ότι δεν υπήρξε έλλειμμα νομιμοποίησης είναι δύσκολο να το πούμε διότι η Τρόικα εκφράζει όργανα νομιμοποιημένα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανεξάρτητα αν έκανε καλά ή κακά που, ήρθε στην, που μπήκε στην Ευρώπη τι προσέφερε, αν ήταν απαραίτητο αλλά είναι ένα όργανο στο οποίο μετέχουν οι χώρες και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι νομοποιημένο όργανο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά οι διαδικασίες δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν έπαιζαν ρόλο, ε, δεν κάναν διαβούλευση, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό σε μια τυπική διαδικασία ανταλλαγής κάποιων απόψεων υπάρχουν κενά αναμφισβήτητα που όλους μας ενοχλούν και μας καλούν να τα αξιολογήσουμε και να τα αναφέρουμε. Ε, η σύνθεση και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ε, είμαστε η το πολιτικό μου κόμμα το πρώτο που κατήγγειλε τη σύνθεση των προγραμμάτων η ισορροπία μεταξύ ε, εσωτερικής υποτίμησης και ε, μεταρρυθμίσεων ή αντιστάσεις και οι δυνατότητες μιας χώρας σαν την ελλάδα αν πάρω παράδειγμα τη χώρα μου να ανταποκριθούν στα χρονικά διαστήματα που επέβαλαν τα προγράμματα όλα αυτά είναι προγράμματα, θέματα προς συζήτηση. αυτή τη στιγμή όμως πρέπει ε, να είμαστε απαιτητικοί διότι τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα έλθουμε στο τέλος αυτών των προγραμμάτων με τον καλύτερο τρόπο για να αποκατασταθεί και η ισορροπία η κοινωνική μέσα στις χώρες και η τρόικα ή οποιοδήποτε πως θα λέγονται ελεκτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται μέσα στο κοινοτικό κεκτημένο. Και όσο για το πρώτο κομμάτι πρέπει να φανεί καθαρά η προσπάθεια που έγινε στις διάφορες χώρες και χαίρομαι που ο Ότμαρ Κάρας έκανε τροπολογίες ο ίδιος για τη χώρα μου αναγνωρίζοντας την πρόοδο στη δημοσιονομική προσαρμογή και στον αριθμό των μεταρρυθμίσεων και το βάθος των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει και πώς όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα ή στην ανεργία, στην έλλειψη ε, ε, αναπτυξιακών ρυθμών, ε, πώς θα ληφθούν υπόψη στην τελευταία αξιολόγηση και επίσης στη βιωσιμότητα του χρέους. Έχουμε μπροστά μας δυνατότητες να διορθωθεί, να αποκατασταθεί αυτή η υστέρηση της επιτυχίας του προγράμματος. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι με μια συλλογική προσπάθεια και πάνω απ' όλα με τις θυσίες των λαών βρισκόμαστε στην επίτευξη του στόχου που είναι το πρωτογενές πλεόνασμα και από εκεί να μπορέσουμε με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς να δούμε την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο χρειάζεται να ασχοληθεί και με το επόμενο βήμα. Είμαστε ένα πολιτικό όργανο, δεν είμαστε ελεγκτικό συνέδριο. Με το, επόμενο βήμα που θα είναι όλη αυτή η πρωτοφανής κατάσταση με τις συνέπειες της τις θετικές και τις αρνητικές πώς θα κεφαλοποιηθεί για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτικές στις χώρες. Και αυτό είναι και το πνεύμα των δικών μου τροπολογιών για να μην αναφέρομαι συγκεκριμένα διότι δεν υπάρχει χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Indeed, uh, σας, σας κατευχαριστούμε κυρία Κράτσα και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Όλε Σμίτ. Εγώ θα είμαι σύντομος η πρόεδρος είπε ότι μερικές χώρες ενδιαφέρονται πιο πολύ από άλλες. Εγώ θα έλεγα ότι όλες οι χώρες, ιδιαίτερα οι έξω από την Ευρωζώνη, πρέπει να καταλάβουν ότι άμα δεν διορθωθούν τα πράγματα τώρα, τότε η χώρα μου δεν θα μπει ποτέ στην Ευρωζώνη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω καλά, σέβομαι πολύ τον κύριο Κάρας και τον κύριο Γκόκ, Εδώ είμαστε σε πολιτικό όργανο, δεν είμαστε τεχνικό όργανο και φυσικά καταλαβαίνω ότι τελικά θα υπάρξει κάποιο συμβιβασμό όπως πάντοτε και εγώ θα ακολουθήσω τον σκιώδημο αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και για μένα που ασχολούμαι με την πολιτική σχεδόν 40 χρόνια η προσωπική και η συλλογική ευθύνη είναι το κλειδί της δημοκρατίας. Καμιά φορά πρέπει κανείς να εκδιωχθεί από την πολιτική του θέση γιατί απέτυχε, γιατί τα έκανε σαλάτα. Και με απογοήτευσε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν παραδέχτηκε κανένα λάθος του. Νομίζω ότι είναι προφανές σε μια δημοκρατία ότι πρέπει κανείς να το κάνει. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε ορισμένους ότι τον Μάιο του 2000 δεχτήκαμε μία έκθεση του Ρόμπερτ Γκέμπελς που έλεγε ότι η Ελλάδα έπρεπε να μπει στην Ευρωζώνη. Μόλις το ξαναδιάβασα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα δεχτήκαμε όλα, όλα. Και η Περβάνς Μπερές ήταν εκεί και ψήφισε, ο Ότμαρ Κάρας ήταν εκεί και το δέχτηκε. Βέρνερ Λάγκεν ήταν εκεί και ψήφισε και ακόμη και ο Σμίτ ήταν εκεί και ψήφισε. Έχουμε ή δεν έχουμε κι εμείς κάποια ευθύνη για όλα αυτά. Εγώ θα έλεγα ναι. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα η κυρία και εμεις Γιατί, για ένα λεπτό όμως γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι συνεισηγητές. Δεν είστε βέβαια μέλος της Επιτροπής, αλλά θα μιλήσετε. Παρακαλώ όμως μόνο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά εκπροσωπώ το λαό της Κύπρου και υπάρχουν αρκετές αναφορές για την περίπτωση της Κύπρου και στη συζήτηση και στην έκθεση. Έχω καταθέσει συνολικά 11 τροπολογίες. Ε, από αυτές θεωρώ σημαντικότερη την 227 τροπολογία, η οποία εξηγά ακριβώ πώς ο καλύτερος μαθητής για ένταξη στην Ευρωζώνη την περίοδο 2004-2008 τελικά βρέθηκε στην ανάγκη να μπει σε μνημόνιο. Δυστυχώς η έκθεση της Κύπρου στην ε, ελληνική οικονομία και τη απόφασης της Ευρωομάδας για διάσωση του ελληνικού δημόσιου χρέου τον Μάιο του 2011 στήχησε στην Κύπρο 4,5 δισεκατομμύρια που ήταν ακριβώς 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας μου. Γι' αυτό η Κύπρος αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια. Δυστυχώ όμω, αντί να έχει κοινοτική αλληλεγγύη ε, δέχτηκε ένα πρωτοφανέ κούρεμα καταθέσεων για το οποίο ο κόσμο τη Κύπρου νιώθει ιδιαίτερα αντικειμένος. Αναμένουμε από αυτή την έκθεση πραγματικά να βγάλει ρεαλιστικά συμπεράσματα. Και η άποψή μα είναι ότι ναι, χάσαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 4,5 δι, ζητήσαμε 5,6 δι και τελικά μα δόθηκαν 10. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Οι μονόπλευρε πολιτικέ λιτότητα χωρί ανάπτυξη και χωρί επενδύσει δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Δεν μπορεί με μια συνταγή για όλους να γίνονται επίλυση προβλημάτων αυτό είναι λάθος και υπάρχουν και δύο μέτρα δυστυχώς και δύο σταθμά διότι είδαμε τη βελγική τράπεζα αντέξια εδώ στις βρυξέλλες να ζητά 100 δισεκατομμύρια γιατί είχε πρόβλημα και να τις δίνονται ενώ στην Κύπρο ζητήθηκε μόνο 5,6 και αυτό ήταν τεράστιο λάθο. Και θα ήθελα ο κύριο Λάγκε επειδή έχει πει ότι εμεί ζητήσαμε το κούρεμα θεωρώ ότι αυτό δεν ήταν σωστό και πρέπει να το τεκμηριώσει. Τελειώνοντα, θεωρώ ότι οι 11 τροπολογίε που έχω θέσει αγγίζουν στον τύπο των ύλων και η θερμή μου παράκληση είναι αυτέ να υιοθετηθούν από την Επιτροπή. Thank you ε, Σας κατευχαριστώ. Το λόγο τώρα οι συνεισηγητές, ο κύριος Κάρας καταρχήν από το ΕΛΚ. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση και επίσης ε, και για το ότι τελικά από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούν για τη μορφή που πρέπει να λάβει η έκθεση. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, προτάσεις σας. Θέλουμε τη στήριξή σας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και παρακαλώ όλους να είναι οι δυνατόν στη διάθεσή μας για να προετοιμάσουμε από κοινού τις συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Καράς. Από τους σοσιαλιστές ο εξηγητής κύριος Γκόκ. Μερικά δυο λόγια για να λήξει αυτή η συζήτηση. Άκουσα με προσοχή όλους και έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι μίλησαν θεωρούν ότι η έκθεση είναι και πολύ λεπτή και πολύ συμβολική και όλοι νομίζω θέλουν το Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια θέση στέναρη πριν δείξει η θητεία του. Διότι είναι το μόνο όργανο που έχει εκλεγεί άμεσα και μπορεί να κάνει προτάσεις για το μέλλον για τον έλεγχο των μηχανισμών που θα ισχύσουν στην οικονομική διακυβέρνηση των χωρών με πρόγραμμα αλλά και γενικότερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι αρκετά ικανοποιημένο. Ο Βέρνερ Λάγκεν μόλις έφυγε, αλλά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί ακόμη και ο Βέρνερ Λάγκεν είπε σήμερα ότι το σχέδιο που είχαμε υποβάλει ήταν εξαιρετική βάση συζήτησης ή εκκίνησης και σε αυτή τη βάση και εμείς ελπίζουμε να πετύχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία. Πολλοί επέμειναν ότι δεν πρέπει να τα πούμε ιδεολογικά, σχεδόν όλοι. Ενδιαφέρον και αστείο αρκετά. Θα σας υπενθυμίσω ότι προηγουμένως υπήρχαν τόσοι ιδεολόγοι υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων όσοι και σκέφτονταν ότι το κράτος είναι το πρόβλημα. Άρα είναι καταμερισμένες επαρκώς οι ευθύνες και οι ιδεολογίες. Πώς να κάνουμε όμως αξιολόγηση, με ποια βάση. Ε, με βάση την πραγματικότητα. Εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με την οικονομία και η πραγματικότητα είναι αριθμή. Ο Ότμαρ είπε πριν ότι οι αριθμοί δεν λένε και πολλά από μόνοι τους. Αλλά οι αριθμοί είναι πεισματάρικοι έξι χρόνια συνεχούς ύφεση στην Ελλάδα, τέσσερα-πέντε χρόνια σε δυο άλλες χώρες με πρόγραμμα, ανάπτυξη που δεν υπάρχει σχεδόν στην Ιρλανδία, χρέωση που ξεπερνάει παντού, ε, τέλος πάντων τα λέω παντού, εννοώ σε τρεις από τέσσερις χώρες άνω του 20% του ε, ακαθάριση του προϊόντος, ε, το κριτήριο που χρησιμοποιεί δηλαδή το Δουνουτού. Άρα αφού υπάρχουν ακόμη οι παράγοντες που δημιούργησαν την κρίση δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες ότι τελείωσε η κρίση και ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν οι αριθμοί και το Δουνουτού μας λέει ότι ο πολλαπλασιαστής είναι γύρω στο 1,5. Όταν δηλαδή ξεκονομούμε 10 ευρώ από τις δημόσιες δαπάνες μειώνεται κατά 15 ευρώ η οικονομία. Αυτό είναι θέμα αντικειμενικό και αυτό οδήγησε την Τρόικα να μειώσει κάπως τις προβλέψεις και τους στόχους της. Ο Λάμπερτ που έφυγε και αυτός σωστά είπε ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Πράγματι και γυναίκες εντάξει, ναι γιατί στα γαλλικά άνθρωπος λέγεται άντρας εντάξει. Ναι, μην με διακόπτετε τώρα για τις γυναίκες και θα καθυστερήσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι και πράγματι είναι ρόλος της Επιτροπής Απασχόλησης να ασχοληθεί με αυτά, αλλά επίσης και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των κοινωνικών συμβάσεων ή μη συμβάσεων πάνω στην οικονομία. Και η Άννα ακριβώς ξέρει ότι στην Πορτογαλία συζητιέται το κοινωνικό συμβόλαιο που ισχύει και το οποίο αρνήθηκε η Τρόικα. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να το θίξουμε. Ποιος θα αποφασίσει για αυτά τους προβλήματα, ας πούμε τις συμφωνίες για τον ελάχιστο μισθό. Αν υπάρχει δυνατότητα συνένεση σε μια δημοκρατική χώρα, έχει το δικαίωμα η Τρόικα να έρθει να μας εξηγήσει ότι δεν θα εφαρμοστεί η συμφωνία ενώ η ίδια η Τρόικα δεν έχει νομικό υπόβαθρο και οι συμφωνίες μεταξύ των εταίρων της δεν δημοσιεύονται πουθενά. Σημερίζομαι και τις ανησυχίες της Σάρων Μπόλς που έφυγε και αυτή προκειμένου για τη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν τα είπε όπως θα τα πω εγώ, αλλά νομίζω ότι το ευρώ είναι το πρόβλημα, όχι η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό τη θητεία είχε. Είχε δικαίωμα λοιπόν να επιβάλλει το bailout της Ιρλανδίας. Είχε εντολή να αποφανθεί για την αναδιάρθρωση μη του ελληνικού χρέους. Όλα αυτά δεν ξέρουμε ποιος και πότε τα αποφάσισε. Και για να το πω πιο ομά, τίθεται εδώ το, το θέμα της δημοκρατίας και εδώ συμφωνώ με τον συνεισηγητή μου. Το κεντρικό θέμα είναι το θέμα της δημοκρατίας και συμφωνούμε 100% όχι μόνο με τον συνεισηγητή, με όλους που μίλησαν σήμερα ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας πρέπει να επεκταθεί και να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με ευρωδημοκρατική διαχείριση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς στο Κοινοβούλιο δημοκρατικά, αλλά μέσω της κοινοτικής μεθόδου. Είτε πρόκειται για τους φιλελεύθερους, για την ΚΟΥ, για οποιαδήποτε ομάδα, όλοι συμφωνούμε ότι μονο η δημοκρατία θα επιτρέψει τη λήψη της απόφασης και τη λύση του προβλήματος για να δούμε ποια ακριβώς πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να φτάσουμε σε πολύ καλό συμβιβασμό εφόσον όλοι είναι επικοδομητικοί και δεν αποδομήσουν ό,τι προσπαθήσαμε να κάνουμε μέχρι τώρα, να ξεπλέξουν το πουλόβερ μας. Είμαι αισιόδοξο και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους και θα συναντήσουμε αύριο τους Σκιώδης για να δεφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκόκ. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά μπορεί να εξεταστούν και δεύτερη φορά οι τροπολογίε στις 20 Φεβρουαρίου, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Μόλις το μάθουμε σίγουρα θα σας το γνωστοποιήσουμε. Στην οίκονη ψηφοφορία θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια τον Μάρτιο. Αύριο στις 9 Αποκινούμε τη Λίμπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.